Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Προτείνω να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, αλλά δεν χρειάζεται να τον ε, κατασπαταλούμε. Οπότε, συνεχίζοντας τις χθεσινές μας συζητήσεις ε, με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ιδρύματα, περνάμε στην απαλλαγή για αυτούς τους οργανισμούς και τα ιδρύματα. Έχουμε κοινή συζήτηση. Θα σας αναφέρω τις διάφορες απαλλαγές με τη σειρά που περιγράφονται στην ημερήσια διάταξη και θα σας ε, σχολιάσω και κάποιες τροπολογίες. Σημείο 13. Πρώτα, απαλλαγή 2012 για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω λάβει τρεις τροπολογίες Με την πρώτη δεν έχω πρόβλημα. Αντίθετα, για τη δεύτερη, ναι μεν χαίρομαι για την επιτυχία που είχαν αυτές ε, οι δειγματοληπτικές ε, συναλλαγές. Ο κύριος Όρη μας προτείνει να περιορίσουμε αυτή τη διαδικασία και να πούμε ότι θα πρέπει να την απλουστεύσουμε. Και η τρίτη τροπολογία αναφέρει ότι οι επιλογές απλουστευμένης απόδοσης δαπανών μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα των λαθών. Αν θέλετε να το συζητήσουμε, εγώ πάντως δεν έχω πιστεί από το επιχείρημα του κυρίου Όρη. Σημείο 14. Απαλλαγή 2012 για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ETF. Μια στιγμή να κάνω ό,τι έκαναν χθες μερικοί συνάδελφοι. s'agissant euh, de ETF. Σημείο 14 λοιπόν. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Έχουν κατατεθεί δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά την παρουσίαση της δημοσιονομικής κατάστασης της 31 Δεκεμβρίου 2012. Ουσιαστικά γίνεται μια υπενθύμηση Ενό γεγονότο που έχει ήδη συμβεί, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και η δεύτερη τροπολογία μιλάει για την έγκαιρη εκκίνηση της διαδικασίας. Δεν έχω πρόβλημα ούτε με τη δεύτερη τροπολογία. Πάντως για το Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουμε ένα πρόβλημα με την περσινή χρονιά, το 2013. Βέβαια τώρα μιλούμε για την απαλλαγή του 2013 11 λέει πρόεδρο, 12 λέει μέρη σε διάταξη. Αλλά αν έχουμε πρόβλημα στο, το 2013 ίσως ε, επαναληφθεί. Θα πρότεινα λοιπόν μια σύντομη προφορική τροπολογία για το Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ε, παράταση της ε, θητείας της κυρίας Σερμπάν. Εγώ χαίρομαι που ανανεώθηκε η σύμβασή της, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτική και αξιοθαύμαστη διευθύντρια, αλλά η διαδικασία της ανανέωσης ε, της θητείας γίνεται με πλήρως αδιαφανή τρόπο, κατά τη γνώμη μας. Και έλαβα μια επιστολή από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, που θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχαν στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβεβαίωσε την ανανέωση της θητείας της κυρίας Σέρμπαν, αλλά όπως ξέρετε η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η κυρία Σάρα Πάρκιν που χθες μίλησε εκτενώς εμποδίζοντας τους ε, ε, υπόλοιπου ε, ευρωβουλευτέ να μιλήσουν γιατί δεν έμεινε χρόνο και δεν είχαμε διερμηνία και μάλιστα ε, έφυγε από τη συνεδρίαση και πριν από το πέρα τη συνεδρίαση και δεν μα ενημέρωσε καν για τη διαδικασία διορισμού. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται ιδιαίτερα και με οριζόντιο τρόπο για την άσκηση των εξουσιών αυτής της, ε, αυτών των υπηρεσιών και ιδρυμάτων. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε να περάσει έτσι το θέμα ασυζητητή. Θα σας υποβάλω μέχρι αύριο το μεσημέρι μια προφορική ερώτηση, γιατί πρέπει να δούμε αυτό το θέμα της απαλλαγής. Α, ψηφίζουμε σήμερα. Εντάξει, θα σας υποβάλω εντός ολίγου προφορική τροπολογία, γιατί πιστεύω ότι το μήνυμα θα πρέπει να περάσει. Σημείο 15 τώρα. Απαλλαγή για τον οργανισμό του Μπιλμπάου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες για την απαλλαγή αυτή και επ' ευκαιρία της απαλλαγής του 2012 θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την έλλειψη νέας στρατηγικής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τηλεγραφικά έρχομαι και στο σημείο 16 που αφορά την απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβιώσεως και Εργασίας. Το Ίδρυμα Eurofound. Εδώ έχουμε αρκετές τροπολογίες, αλλά κανένα πρόβλημα γιατί είναι υπέρ και των 8 τροπολογιών. Αλλά παρόλα αυτά θα τη σχολιάσω. Η πρώτη τροπολογία είναι του κυρίου Σέρτζο Γκουτιέρες Πριέτο, που θέλει να αναφέρουμε το Eurofound και όχι το Ίδρυμα απλώς. Δεύτερη τροπολογία της κυρίας Χάρκιν. μας υπεθυμίζει το πλαίσιο που δικαιολογεί την επιδείνωση των συνθήκων σε ορισμένα κράτη-μέλη. Τροπολογία 3 του Σέρτζιο Κουτιέρες είναι ουσιαστικά μια επανάληψη της πρώτης τροπολογίας, δηλαδή αντικαθιστά το, το Ίδρυμα από το Eurofound. Το ίδιο και η τροπολογία 4. Δεν έχω πρόβλημα. Τροπολογία 5 της κυρίας Χάρκιν. Η κυρία Χάρκιν λέει στην πέμπτη τροπολογία ότι υπενθυμίζοντας την ικανοποίηση για το ελεκτικό συνέδριο που χαρακτήρισε νόμες και κανονικές υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών, για το οικονομικό έτος 2012. Η κυρία Χάρκιν ε, προτείνει ε, να επισημάνουμε ότι παρουσιάζεται με σαφήνεια η δημοσιονομική κατάσταση 31 Δεκεμβρίου 2012. Συμφωνώ κι εγώ. Τροπολογία 6. Τσάμπα όρη. Ο κύριος Όρη αναφέρει ότι στον τίτλο 1 και 2 ελήφθησαν διορθωτικά, μέτρα για τις δηλωθήσεις καταγγελίες το προηγούμενο έτος. Κανένα πρόβλημα. Τροπολογία 7. Σέρτζο Κουτιέρες Πριέτο. Επαναλαμβάνει επίσης, όπως και στις προηγούμενες, ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να αντικατασταθεί από το Eurofound. Και τροπολογία 8 το ίδιο αναφέρει. Προσθέτει όμως ένα σχόλιο που λέει ότι όλες οι συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου σχετικά με τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης έχουν εφαρμοστεί σφαιρικά. Συμφωνώ και με την τροπολογία 8 λοιπόν. Δέχομαι και τις 8 τροπολογίες και τελειώσαμε με το Eurofound. Περνάμε στο 17. Την απαλλαγή για το Σεντεφόπ. Εδώ έχουμε τρεις τροπολογίες. Η πρώτη είναι της κυρίας Χάρκιν που ουσιαστικά είναι αντανάκλαση της αντίστοιχης τροπολογίας για το Eurofound. Εκεί θυμίζει ότι απαιτούνται νέοι μέθοδοι κατάρτισης ε, την εποχή που διανύουμε. Τροπολογία 2 είναι παρόμοια με αυτή που είχε καταθέσει η κυρία Χάρκιν για το Eurofound. Υπενθυμίζει ότι παρουσιάστηκε με σαφήνεια η δημοσιονομική κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ενώ η τροπολογία 3 του κυρίου Τσάβα Όρη λυπάται για το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη διορθωθεί ικανοποιητικά τα εντοπιστέντα ελλείμματα του προηγούμενου έτους. Και δεν συμφωνώ, γιατί έγινε μια ανανέωση του προσωπικού. Στο 18, που αφορά όλες τις ε, υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδρύματα, έχουμε τέσσερις τροπολογίες. Η πρώτη είναι του κ. Τσαμπαόρη, κανένα πρόβλημα. Και μετά έχουμε τρεις τροπολογίες για την ίδια παράγραφο, την παράγραφο 3. Οι τροπολογίες είναι του κυρίου Πριέτο, του κυρίου Όρη και της κυρίας Χάρκιν. Θα σας πρότεινα μια συμβαστική τροπολογία που καλύπτει και τις τρεις και που επιμένει στη σημασία που έχει η συνεργασία μεταξύ των ε, οργανισμών. Τις παρακινούμε να συνεχίσουν τις προσπάθειες για καλύτερη συνεργασία η συνεργασία αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σχέδιο δράσης, τα ερευνητικά προγράμματα, την κατάρτιση ερευνητικών ε, σχεδίων και τις μεθόδους παρατήρησης. Επίσης, αυτή η συνεργασία θα πρέπει να έχει απτά αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν. Ολοκλήρωσα την παρουσίασή μου. Το νέο στοιχείο είναι δεδομένη κατάστασης στο Ίδρυμα επαγγελματική εκπαίδευση. θα πρέπει να κάνουμε υποβάλουμε κάποιες παρατηρήσεις για την ανανέωση της θητεία και της κυρίας Σέρμπαν. Βέβαια θα βάζουμε ιδιαίτερα την διευθύντρια αυτή, είναι αξιοθαύμαστη και αυτή παρατηρείται δεν έχει καμία σχέση με το πρόσωπό της. Είναι θέμα της διαδικασίας ανανέωσης που είναι διαφανής. Ευχαριστώ και ο λόγος των Αλεχάνδρο Σέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς για το Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα ήθελα να μιλήσω, το ETF. Είναι σαφέστατα αυτά που μας είπατε και θα υπερψηφίσουμε την προφορική σας τροπολογία, αλλά θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια για να αποφευθούν οι παρεξηγήσεις, ώστε να μην εκλειφθεί η δυσαρέσκειά μας ως προς τη διαδικασία με ένα είδος μοφής προς το πρόσωπο της κυρίας Σέρμπαν. Γιατί το τονίσατε κι εσείς, αλλά θα ήθελα να το επισημάνω κι εγώ για να γίνει πλήρης διαχωρισμός της ουσίας από τη διαδικασία. Γιατί ε, θεωρούμε ιδιαίτερα αξιόλογη την Διευθύντρια. Η παρατήρησή μας αφορά μόνο τη διαδικασία ανανέωσης της θητείας της. Ο κύριος Όρη. Εγώ θέλω να παρέμβω μόνο σύντομα όσον αφορά την εκτέλεση του Γενικού Προϋπολογισμού της ε, χρήσης 2012. Εάν κατάλαβα καλά, Πρόεδρε, εσείς ερμηνεύσατε την τροπολογία μου, την υπαριθμό 3, που αναφέρεται στη νέα παράγραφο 6 και συγκεκριμένα το δεύτερο τμήμα αυτής, σύμφωνα με την οποία οι κανόνες θα πολλαπλασιάζονται. Εγώ δεν το λέω αυτό. Εγώ λέω ότι εντάξει η απλοποιημένη διαδικασία. Ωστόσο, αυτό σημαίνει πως ορισμένες λεπτομέρειες δεν θα τις γνωρίζουμε και ότι αν υπάρξει κάποιο σφάλμα δεν θα μπορούμε να το εντοπίσουμε. Δεν σημαίνει αυτό ότι αυξάνονται τα σφάλματα. Λέω απλά ότι με την απλοποιημένη διαδικασία και διακόπτει ο μιλητής. Υπάρχει εκπρόσωπος της Επιτροπής που θέλει να παρέμβει. μα δεν είχα ολοκληρώσει. Περίμενα να τελειώσετε με μεταξύ σας ε, διαβούλευση. Περίμενα να με ακούσετε. Ε, ναι, έχετε δίκιο έχετε ίσως την εντύπωση ότι δεν σας άκουγα με τόσο πολύ προσοχή. Λοιπόν, τώρα είμαι όλη αυτιά και έχετε και πάλι το λόγο. Παναλαμβάνω. Εγώ δεν θέλω να πω ότι λόγω αυτής της απλοποιημένης διαδικασίας ε, ε, ε, θα αυξηθούν τα σφάλματα ή οι παρατυπίες αλλά ότι εάν υπάρξουν παρατυπίες δεν θα είναι τόσο εύκολο να εντοπιστούν γιατί έχουμε και πιο περιορισμένο χρόνο και δεν θα καταφέρουμε να μελετήσουμε τις λεπτομέρειες. Ίσως η Κομισιόν λόγω μεγαλύτερου συντονισμού να, μην, να θεωρεί ότι δεν χρειάζονται όλες αυτές οι λεπτομέρειες οπότε ε, εγώ μπορώ και να το δεχτώ απλά ήθελα να εκφράσω ποιο είναι το πρόβλημά μου. Μάλιστα. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Κομισιόν. Ίσως ε, να δούμε πώς ε, θα αντιδράσει, πόσο πρόκειται για διαδικασίες ε, διορισμών ε, το 2 και το 3. Τα δύο συνδέονται. Η Κομισιόν λοιπόν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς θα θέλαμε να σχολιάσουμε όλες ιδιαίτερως αυτά, αυτές τις τροπολογίες όσον αφορά την χρήση απλοποιημένων διαδικασιών και να τονίσουμε ότι μετά από προηγούμενες διαδικασίες και συστάσεις μάλλον απαλλαγή από την Επιτροπή σας, έχουμε επενδύσει σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών για την απλοποίηση, στην απλοποίηση, για να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο και το ποσοστό σφάλματος. Επίσης έχουμε προωθήσει την απλοποίηση στην ε, τρέχουσα περίοδο. Αυτό σημαίνει ενίσχυση των απλοποιημένων διαδικασιών και πράγμα το οποίο θα συνεχιστεί και κατά την περίοδο 2014-2020 τα αποτελέσματα έχουν επιβεβαιωθεί σαφώς στην έκθεση ε, ε του 2012 όπου τονίζεται ότι όχι μόνο το αποτέλεσμα ήταν η μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά υπήρξε αντίκτυπος και στο περιθώριο σφάλματος, μάλλον στα σφάλματα που μειώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό και θεωρούμε πως αν αυτή η τροπολογία διατηρηθεί, θα υποβαθμίσει ε, την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Ε, τώρα, σε σχέση με το ETF, θεωρούμε πως... Ε, Δεν, είναι, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε εδώ για αυτόν τον ε, διορισμό. Euh, Μάλιστα, σας ευχαριστώ για αυτές τις ευκρινήσεις. Εγώ προτείνω, αγαπητέ συνάδελφοι Φεόρη, Εγώ πιστεύω πως όταν μπορούμε να απλοποιήσουμε ε, δεν νομίζω πως μπορεί η Κομισιόν εδώ να θεωρηθεί υποπτή είτε είναι για την ιδέα είτε είναι για τις, τους οργανισμούς ή να κατηγορηθεί για ελαφρότητα σε θέματα ελέγχου και υποπτία της διαδικασίας ε, χρήσης των, του δημόσιου χρήματος. Όλοι οι φορείς επιμένουμε πάντοτε για να πηγαίνουμε προς διαδικασίες πιο απλοποιημένες από τη στιγμή που δεν αυξάνεται ο κίνδυνος ατασταλίας ή κακοδιαχείρισης. Και εδώ το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο είναι αυτό που λέει ότι αυτές οι, προπημένε οι διαδικασίες επιτρέπουν την μείωση των διοικητικών κινδύνων. Εγώ θέλω να βασιστούμε λοιπόν σε αυτή την παρατήρηση του, του ελεγκτικού συνεδρίου που είναι απόλυτα θετική κατά τη γνώμη μου και ήταν και το νόημα του δεύτερου τμήματος της παραγράφου 6 της τροπολογίας μας. Παράγραφος 6 που θέλαμε να καταργήσουμε, πράγμα που θέλετε μάλλον να καταργήσουμε, πράγμα που θα ήταν κρίμα. Εγώ προτείνω λοιπόν να αποσύρετε την τροπολογία 2 και αντιθέτως στη 3 να τροποποιήσετε κάπως το κείμενο έτσι ώστε να διατηρηθεί το πνεύμα επαγρύπνησης σε σχέση με τους κινδύνους κακής εφαρμογής. Αλλά κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε λίγο πίσω στα όσα επίσημα προτείνονται στην τροπολογία 3. Ελπίζω να με καταλάβατε. Και ότι στο τέλος αυτής της συζήτησης θα έχουμε νέες προτάσεις ώστε να συνεχίσουμε στο πνεύμα συνεργασίας που είχαμε ανέκαθεν ναι, γύρω από αυτά τα δημοσιονομικά ε, θέματα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτά τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Και θα ψηφίσουμε, θα ξανασυζητήσουμε στις 12 Φεβρουαρίου και ε, Ελπίζω πως θα μπορέσουμε και προφορικά να συζητήσουμε για τους διορισμούς και ελπίζω και ότι ο Τσάμπα Όρη θα μπορέσει να κινηθεί κάπως, να μετακινηθεί κάπως από τις θέσεις του για αυτή τη διαδικασία ε, και ο έλεγχος προπολογισμού ψηφίζει στις 17 Μαρτίου. Οπότε λοιπόν, έχουμε χρόνο, το ολοκληρώσαμε τώρα αυτό το κομμάτι της σημερινής διέταξης. είναι 9 και 34 και προβλέπεται να περάσουμε στο σημείο 20, δηλαδή στις ψηφοφορίες για την έκθεση πρωτοβουλίας που μας επιτρέπει να κάνουμε συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, την απασχόληση κοινωνικές πτυχές μέσα στο πλαίσιο της, του έτους ανάκαμψης 2014. Πρόκειται για την έκθεση Πρόκειται για την έκθεση του κυρίου Γκουτιέρες Πριέτο. Alors, euh, Ωραία λοιπόν. Αντιμετωπίζουμε βέβαια μία μικρή δυσκολία την οποία σας επισημαίνω. Πρώτον, έχετε όλες και όλοι τις κάρτες σας. Ποιος ή ποια δεν έχει. Μία σοσιαλίστρια. Τέλος πάντων, δεν είναι και παραπάνω η ψήφη, αλλά δεν έχει κάρτα. Τώρα, η δυσκολία που έχουμε είναι Φαίνεται πως οι συμβιβασμοί ήταν περίπλοκοι, οι διαπραγματεύσεις μακρές και φαίνεται πως ορισμένες ρυθμίσεις για τους συμβιβασμούς έγιναν εκπρόθεσμα. Και επομένως αυτές οι προσαρμογές δεν εμφανίζονται στα κείμενα που έχουν περιληφθεί στην λίστα ψηφοφορίας αφενός και όλες οι πολιτικές ομάδες δεν έχουν λάβει γνώση οι κανόνες που σταθερά βρίσκουν εφαρμογή σχετικά με τις λίστες ε, ψηφοφορίας εδώ και που εντάσσονται σε μια μεθοδολογία εργασίας την οποία ενέκριναν οι συντονιστές στις αρχές της θητείας και όπου οφείλουμε να την σεβαστούμε εάν θέλουμε να εργαστούμε υπό καλές συνθήκες. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσαρμόσουμε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες όταν θα ε, εκφωνούνται, αλλά βέβαια αυτό κάνει την δουλειά όλων μας πιο δύσκολη. Αυτές οι δυσκολίες τώρα, λοιπόν, που ανέφερα, αναφέρω στο Q, Q δηλαδή, R, O, O, επίσης στην 81 και 129, οι οποίες έχουν αποσυρθεί όμως. Αν λοιπόν δεν έχετε αντίρρηση να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Πριν από την παράγραφο 1 έχω τη συμβαστική Ι τεσσάρων ομάδων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από την συμβαστική τροπολογία η 61. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Παράγραφος 2. J. Συμβαστική J. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Παράγραφος 3. Συμβαστική κάπα τριών ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. Παράγραφος 4. 75 Φιλίπ Μπάκερ που ε, επιδιώκει διαγραφή για τις 76 και 77 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κυρία Εσαγιά, αν ψηφίσετε κατά, θα μπορέσετε να ψηφίσετε τροπολογία σας. Ψηφίσατε όλες και όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. 19 υπέρ 18 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία DeBacker, που σημαίνει ότι οι τροπολογίες 76 και 77 εκπίπτουν. Παράγραφος 5, 2 ταυτόσιμες τροπολογίες 78 και 79. DeBacker, Εσαγιά. Τις ψηφίζουμε. Και αυτέ επιδιώκουν την διαγραφή Είπε. Α, με συγχωρείτε, διακόπτη πρόεδρος. Δεν υπάρχει, ε, δυστυχώς, δεν ακούω διερμηνία από τα φιλανδικά, κύριε Πρόεδρε. Κατάλαβα, κατάλαβα, ναι, λέει η Πρόεδρος. Μια στιγμή Υπάρχουν τα φιλανδικά, υπάρχουν τα φιλανδικά. Κανονικά θα πρέπει να έχετε. Ναι, τώρα μάλιστα, τώρα του ακούω. Καλά. Γι' αυτό δεν κατάλαβα τι μοίρα επιφυλάξατε στις ε, τροπολογίε μου. Εγώ έλεγα προηγουμένω ότι αν καταψηφίσετε, μάλλον αν υπερψηφίσετε την 75, τότε θα ε, εκπέσει η δική σα τροπολογία η παθημόνη 77. Τώρα επανερχόμαστε όμω, αυτό έγινε, στην 79 που είναι ταυτόσιμη με την 78. Τροπολογία λοιπόν 78 και 79 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ναι, διακόπτει ο διακόπτει πρόεδρος. Για βάλτε το μικρόφωνο σας κύριε Σέρκας. Ε, έχουμε μία ψήφο χωρίς κάρτα, ε, σοσιαλίστρια. Ναι, ναι, ναι, ήταν 19-17, αλλά βάλαμε εμείς 19-18, δηλαδή την υπολογίσαμε. Α, έχω όμως ήδη τώρα την κάρτα μου. Α, πολύ ωραία. Άρα το θέμα ρυθμίστηκε και ευχαριστώ για την πληροφορία. Και συνεχίζω τώρα, λέει η πρόεδρος. Έχει εκπέσει παριθμόν 80. Για την ε, παράγραφο 6 ψηφίζουμε. Α, μια στιγμή. 81. Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ έχει αποσυρθεί. Άρα μπορούμε να ψηφίσουμε την συμβαστική μη, όπως Μιχαήλ, τεσσάρων ομάδων. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Μη παραδεκτή. Πάμε λοιπόν στην ε, τροπολογία 7, η οποία επίσης είναι μη παραδεκτή. Παράγραφος 8. Συμβαστική νη, όπως Νικόλαος, δύο πολιτικών ομάδων με α, που είναι προφορική τροπολογία. Γνωρίζετε όλη την συμβαστική νη. Πολύ ωραία λοιπόν τη θέτω ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Απογιάζει. Νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ας ε, παληθεύσαμε. Νι, όπως Νικόλαος. Ψηφίσατε. 19 ψηφί περ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Άρα θέτω σε ψηφοφορία Το αρχικό κείμενο λοιπόν τότε με την προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ κατά θα επαναλάβω, είπαμε είναι λίγο περίπλοκο. Είχαμε μια συμβαστική τροπολογία νη που είχε σκοπό να διορθώσει μια προφορική τροπολογία επί του αρχικού κειμένου. Αυτή η συμβαστική τροπολογία ωστόσο απερίφθη. Τώρα, Θέτω σε ψηφοφορία λοιπόν την αρχική παράγραφο με την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 88 έχει αποσυρθεί. Παράγραφος, 9. Συμβαστική τροπολογία όμικρον τριών ομάδων. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10, τροπολογία 92 της κυρίας Κρίσλευσκα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ο 93 συμβατή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κύριε Ισηγητά, επιθυμείτε να παρέμβετε. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Αλλά όταν ψηφίσαμε το αρχικό κείμενο της συμβαστικής τροπολογίας ΝΗ, είχαμε κάποιες ε, αλλαγές στη θέση κάποιων ε, συναδέλφων. Θα ήθελα να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί ήταν πολύ ωριακό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε τελικά το αρχικό κείμενο. Μπορείτε να το ελέγξετε. Por ejemplo, Μερικοί ευρωβουλευτέ του ΕΛΚ ήξερα ότι ήταν υπέρ του αρχικού κειμένου και ψήφισαν κατά τι ε, προφορικέ τροπολογίε. Χωρί όμω ε, την ε, τροπολογία δεν είναι δυνατό να... δεν είναι παραδεκτό το αρχικό κείμενο. Παράγραφο 11, 95 της Κυριακονίας υπέρ εγκρίνεται. 94 κρίτης Λευσκά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 12 Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή παράγραφος 13 μη παραδεκτή το ίδιο και η 112 του κυρίου Ντεμπάκερ τώρα υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 103. 103. Ψηφίσατε. Λήξη. Εγκρίνεται με ψήφους 21 υπέρ και 19 κατά. Παράγραφος 15, 104 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105, 106, 107 Εσαϊά, Χάρκιν, Βερονικά Λόπετ, Σαβόρη. Υπέρ, κατά, αποχές. Επαλήθευση, νομίζω ότι απορρίπτονται. Λήξη υπέρ 21 ψήφι κατά 19 εγκρίνεται η 108 εκπίπτει παράγραφος 16 α μια στιγμή η 108 συγγνώμη 108 είναι συμβατή άρα την ψηφίζουμε ψήφι υπέρ της 108 κατά αποχές απορρίπτεται 109 στην παράγραφο 16 διαγραφής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 Κορνέλισεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 17 111 Ντεμπάκερ διαγραφής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 18 στην παράγραφο 18 θα ψηφίσετε πρώτα την συμβαστική Q τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά από την παράγραφο 19, 118 τροπολογία της κυρίας Κορνέλησεν. Θα ψηφίσουμε το πρώτο μέρος μόνο, μα το δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα κάνουμε όμως, συγγνώμη, νομίζω ότι γίνεται επαλήθευση. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Λήξη. 16 υπέρ, 22 κατά, 0 αποχές. Απορρίπτεται και δει Παράγραφο 20. Τροπολογία 120. Δεμπάκερ. Η είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Λέτε να επαληθεύσουμε. Ωραία. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Λήξη. 22 υπέρ, 18 κατά. Έγκρινεται λοιπόν πράγματι. 119 σάρια σαγιά είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι είναι το ίδιο αποτέλεσμα άρα εγκρίνεται παράγραφος 21 συμβαστική R ρο που έχει τροποποιηθεί Ας δώσουμε το λόγο στον εισηγητή που θα εξηγήσει την τροποποίηση της τροπολογίας που έχει προτείνει. Sí, Presidenta, habíamos Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν θυμάμαι καλά, εκεί που μιλούμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τα κράτη-μέλη, λέμε σύμφωνα με τις ε, αντίστοιχες ε, αρμοδιότητές τους. Δεν υπάρχει άλλη αλλαγή. Απλώς παρακινούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να προτείνουν μέτρα κτλ. ανάλογα ή σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Μόνο αυτή η προσθήκη, τίποτα άλλο. Ε, Η πρόεδρος Μπέρες. Στο τέλος εδώ του συμβασμού, μιλούμε για την παράγραφο 21, Ένα λεπτό να διαβουλευτώ και θα επανέλθω. Señora Presidenta, Presidenta, okay. sí, nos dicen... Σουτ, λέει ο πρόεδρος Μπερές. Τροπολογία R, ρο. Θα διαβάσω το κείμενο ως το έχω μπροστά μου και θα μου πείτε τι θα αλλάξετε. Συμβαστική τροπολογία R. Σημειώνει ότι αξιοπρεπείς θέσεις και μισθοί είναι σημαντική και για την κοινωνική συνοχή και για τη δικαιοσύνη μέσα στην κοινωνία, αλλά και για να διατηρηθεί μια ισχυρή οικονομία. Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές των, να προτείνουν μέτρα τα οποία θα αντιμετωπίσουν την ε, ανισότητα στην αξιοπρεπή αμοιβή της εργασίας. Ασκώντας, ασκώντας πολιτικές εργασίας που θα επιτρέψουν να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Τι θέλετε να αλλάξετε σε αυτά τα λόγια. Η παράγραφος είναι τέλεια και μάλιστα είναι η συμβαστική λύση την οποία συμφωνήσαμε με όλες τις πολιτικές ομάδες. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Καμία. Καλά λοιπόν. Χαίρομαι που μπορούμε να ψηφίσουμε την τροπολογία ως έχει ψήφι υπέρ της τροπολογίας ρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία. Άρα εκπίπτουν ορισμένες τροπολογίες και μετά από την 21 ερχόμαστε στην 125 τροπολογία της κυρίας Ιωάννας Κρίσλευσκα. Εισηγητής υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Ε, παράγραφος 22, τροπολογία 126 Ψηφίζουμε ωστόσο απευθεία την σίγμα τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές επαλήθευση, επαλήθευση για την συμβαστική τροπολογία S σίγμα δηλαδή. Ψηφίσατε όλες και όλοι παρακαλώ. 24 ψήφοι υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται και χωρίς αποχές. μετά ένας μεγάλος αριθμός μη παραδεκτών εκτός από την 23 παράγραφο 130 του κ. Ντεπάκερ, ψηφίζεται αυτή υπέρ δικιά ναι, σας είναι υπέρ της 130 λοιπόν κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 29, τροπολογία 141, της κυρίας Λόπε Φοντανιέ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 30, τροπολογία 143, κύριο Ντεπάκρη, υπέρ, κατά, αποχές, μια στιγμή, απορρίπτεται. 142 εκπίπτει, Παράγραφος 31. Διακόπτει η πρόεδρο Μπερές. 144 τεπάκερ υπέρ. Α, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Ναι, για μια στιγμή δεν κατάλαβα τι είχε γίνει. 142 της κυρίας Φοντανιέ, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Ε, ευτυχώς επαγρυπνείται. 31, 144, Φιλίπ Τεμπάκερ, κατά αποχές, Απορρίπτεται. 145. Λόπε Φοντανιέ. Συμβατή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράφος 32. 146. Δεμπάκερ, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 148. Ινές Κριστίνα Ζούμπερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147. Χάιντς Μπέκερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 33, δύο τροπολογίες διαγραφής, 149 και 150, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34, 151, Ρέγνερ, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 35, συμβαστική ταφ, τεσσάρων ομάδων, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά την 35, 155 μπέκερ υπέρ, κατά αποχές, υπέρ, 155 υπέρ, κατά αποχές, σαφώς εγκρίνεται. 156 του ίδιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 36, 157 Φιλίπ Τεμπάκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή αυτή 159 συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 37 συμβαστική γιου τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 38 συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 39, 165, τροπολογία διαγραφής Τεμπάκερ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική FF, δύο μάλλον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράφος 40. 168 διαγραφή Τεμπάκερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. W τώρα τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160, 171 μάλλον έχει αποσυρθεί. 41. Χ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την 41. 173. Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 42. 174. Ρέγνερ υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 21 υπέρ, 18 κατά. Απορρίπτεται. 175. Ναι, ναι, ναι. Έχω δίκιο. Εγκρίνεται λοιπόν, σαφώς. 175. Ζούμπερ, υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. Παράγραφο 43, 176 του Λαϊκού Κόμματος, διαγραφής, υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 177 είναι μη παραδεκτή. Παράγραφο 44. Τροπολογία 178 διαγραφής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική GG, δύο ομάδων, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πολλές μη παραδέκτες. Προχωρούμε στο Y, στην παράγραφο 47, τεσσάρων ομάδων, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυτή. Παράγραφος 49, 189, δεμπάκερ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 188, Λόπε Φοντανιέ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 190 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Παράγραφος 51 Συμβαστική Ζ τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52, 195 τεμπάκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση, επαλήθευση, 195. Ψηφίσατε, λήξη. 22-17, εγκρίνεται εκπίπτει 196, το ίδιο και 194. Μετά 52, 197 Λόπε Φοντανιέ και όροι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 53, όχι, ναι, ναι. Τροπολογία 198 της ίδιας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή. Τροπολογία 199 συμβατή με την 198 την θέτω σε ψηφοφορία τέλο πάντων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 200 εκπίπτει μετά από την 53 έχουμε τώρα Α, συγγνώμη. Μπορούμε να ψηφίσουμε τη 200. Δεν καταπίπτει, άλλωστε ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 53 έχουμε την τροπολογία 201 που πάκι. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Μετά την 53 επίσης συμβαστική τροπολογία ΑΑ από δύο πολιτικές ομάδες. Και εδώ έγιναν κάποιες αλλαγές ε, τη τελευταία στιγμή. Παρακαλώ ο εισηγητής σας μας δώσει τα φώτα του. Στο κείμενο της ε, συμβαστικής τροπολογίας ξεχάσαμε τον όρο consequences, ε, συνέπειες. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτή η παράληψη, αλλά λείπει ο όρος συνέπειες. Λείπει η λέξη συνέπειες από το κείμενο της συμβαστικής τροπολογίας. Δεν ξέρω που χάθηκε. Οπότε το κείμενο λέει, τονίζει ότι τα κράτη-μέλη που δεν εφάρμοσαν σταδιακά τις μεταρρυθμίσεις μπορούν σε μεταγενέστερο στάδιο να βρεθούν σε μια κατάσταση που θα χρειαστεί να επιβάλλουν ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις δραματικές με σημαντικές κοινωνικές συνέπειες. Προσθέτουμε εδώ το συνέπειες Πρόκειται άλλωστε για μια προσθήκη που δεν τροποποιεί την ουσία της συμβαστικής ε, τροπολογίας ΑΑ που ε, τη στηρίζουν τρεις ομάδες. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία ΑΑ. Περνάμε στην παράγραφο 56 και τη συμβαστική τροπολογία ΒΒ από τρεις ομάδες. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 56 έχουμε την τροπολογία 211. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 57. Συμβαστική τροπολογία CC υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για την παράγραφο 58 έχουμε δύο τροπολογίες διαγραφής, 215-216. Σάι Αντεμπάκερ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Παράγραφος 59, τροπολογία 207, Σαρία Σάια. Ζητά διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, αλλά νομίζω ότι εγκρίνεται η ψηφοφορία 217. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ και 16 κατά. Οπότε διαγράφεται η παράγραφος 59. Μετά την παράγραφο 59 που δεν υπάρχει πια έχουμε τη 220 του Μπέκερ. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 Χάιντ Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 222 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 του ίδιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 224 της κυρίας Κορνέλησεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 60. Τροπολογία 225. Σάρια Σάια. Ζητή διαγραφή Ποιος είναι υπέρ της 225, σχετίζεται με τη συμβαστική HH. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε την HH από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 230 της ε, Ινέ Ζουμπέρ. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 229 για την παραγράφα 61 υπέρ κατά αποχές Ποιος είναι υπέρ της 229 της κυρίας Κορνέλησεν κατά αποχές απορρίπτεται. Για το θεωρώντας, μετά το 17 θεωρώντας, τροπολογία είναι υπέρ, backer. κατά αποχές εγκρίνεται. Για την αιτιολογική σκέψη α, τροπολογία 2, backer, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3, καταπίπτει. 4 δε χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 αποσύρεται, μη παραδεκτή. Για την αιτιολογική σκέψη Β έχουμε τη συμβαστική Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από τέσσερι ομάδε ήταν αυτή. Για τη αιτιολογική σκέψη Σ έχουμε τη συμβαστική τροπολογία Β από τέσσερι ομάδε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την αιτιολογική σκέψη Δ έχουμε την τροπολογία 13 εσάια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ε για το αρχικό κείμενο. Προφορική τροπολογία του εισηγητού προκειμένου να γίνει παραδεκτή συμβαστική τροπολογία ε, η ιδεολογική σκέψη μάλλον ε. Οπότε ψηφίζουμε την ιδεολογική σκέψη ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη F. Τροπολογία 16. Ντεμπάκερ. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Επιστρέφουμε στην τροπολογία 15. Κορνέλισεν. Γιατί είναι συμβατή με την προφορική τροπολογία και το αρχικό κείμενο της αιτιολογικής σκέψης ε. Ποιος είναι υπέρ της 15. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 και 18 Εσάια και Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ και Τσάπα Ορή Πανομοιότυπες και είναι υπέρ αφορούν την αιτιολογική σκέψη F Κατά αποχές εγκρίνονται Η 21 καταπίπτει Μετά το F έχουμε την τροπολογία 19 Φωντανιά και όρη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 των ιδίων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Για το G, τροπολογία 22, The Bucker, θέλει τη διαγραφή της του πρώτου τμήματος της αιτιολογικής σκέψης G, γιατί το δεύτερο τμήμα ούτως ή άλλως είναι μη παραδεκτό. Αν ευοδοθεί 22 δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την συμβαστική ΣΕ που την έχει υποστηρίξει και η ομάδα. Το ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 22. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία 22, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία ΣΕ από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το G έχουμε τη συμβαστική τροπολογία Δ από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάλι μετά το G έχουμε την τροπολογία 29, ολοπεφωτανιά και όρη. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η αιτιολογική σκέψη H είναι μη παραδεκτή. Περνάμε στην επόμενη την I. Τροπολογία 38, Debacker ζητά διαγραφή της σχετικής αιτιολογικής σκέψη, οπότε θα ψηφίσουμε αν υπερψηφιστεί την ε. Ποιος είναι υπέρ της 38, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία ε από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη M, τροπολογία 44, χάρκιν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία GG για το ΕΝΗ, αιτιολογική σκέψη από τέσσερι ομάδε, υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία, α, συγγνώμη, τροπολογία 49, υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται του κ. Ντεμπάκερ για την αιτιολογική σκέψη όμικρον. Αιτιολογική σκέψη Π, τροπολογία 54, Σάρια Σάια, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Συμβατή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για την τελική σκέψη Q. Τροπολογία 58. Ζούμπερ. Υπέρ. Για το, οι φιλελεύθεροι μαζί με τους σοσιαλιστές. Αποκλείεται να κερδίσει το ΕΛΚ. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 58. Της κυρία Ζουμπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εδώ ψήφισαν ε, με το ΕΛΚ οι φιλελεύθεροι, οπότε πέρασε η θέση του ΕΛΚ. Τροπολογία 57. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56. είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Συνέζουμπερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά το ρο, τροπολογία 60, Κορνέλησεν. υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Για το παράρτημα, τροπολογία 232, Εσάια, ζητά διαγραφή ολόκληρου του παραρτήματος, ποιος είναι υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Συστάσεις τώρα, τροπολογία 231, δηλαδή 233, συγγνώμη, δηλαδή διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, οπότε ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία II από δύο ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερη σύσταση, 234, 237 αντεμπάκερ. ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε το JJ από δύο ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. 239 ντεμπάκερ. Ζητά διαγραφή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ΚΚ. Από δύο ομάδε. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Σύσταση 4. Τροπολογία 246 ντεμπάκερ. Ζητά διαγραφή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία ΕΕ. Ζήτησε το λόγο εισηγητής για να μας εξηγήσει τι ακριβώς θέλει να ψηφίσουμε. Perdona, Ε, Συγγνώμη. Έχω τον έλεγχο τη κατάσταση. αφήστε τα όλα πάνω μου. Έξι γραμμέ πριν από το τέλος. Αντί απαραίτητο περιθώριο ελιγμών αυξάνουν τους μισθούς. Οπότε θα πούμε θα μπορούσαν να αυξήσουν τους μισθούς. Από εκεί που λέμε αυξάνουν τους μισθούς. Διορθώστε με αν κάνω λάθος ή αν παρεξήγησα την προφορική τροπολογία, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν κάνω λάθο. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία ΕΕ με αυτή τη μικρή αλλαγή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Παράγραφος 4. Παράγραφος 6. Σύσταση 4 Συμβαστική τροπολογία λάμδα λάμδα. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, αν και μάλλον απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 21 ψήφι κατά, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 250 Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ Alors, euh, dans la créativité. Πρώτα θα πρέπει να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία του εισηγητού για το αρχικό κείμενο, τη δημιουργικότητα που μας χαρακτηρίζει σήμερα. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία για το αρχικό κείμενο υπέρ δεν έχουμε πια προφορική. 250. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχέ. Ηλεκτρονικός έλεγχο για την τροπολογία 250. Λόπε Φοντανιέ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος η γυμναστική. Ψηφίσατε όλοι. 19 υπέρ, 20 κατά. Μία αποχή απορρίπτεται. Οπότε πάει παράγραφος 6, γιατί το αρχικό κείμενο δεν ήταν παραδεκτό. Συμφωνείτε όλοι, μάλιστα. Παράγραφος 7. Τροπολογία 251 Ινές Ζουμπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για την σύσταση 5 έχουμε την 252 debugger για διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ. Α, συγγνώμη, λάθος. Η σύσταση 5 είναι μη παραδεκτή, οπότε δεν χρειάζεται καν να ψηφίσουμε τη 252 του κύριου Ντεμπάκερ που ζητά διαγραφή. Το κείμενο είναι ούτως ή άλλως μη παραδεκτό. Περνάμε στην σύσταση 6. Και εδώ έχουμε 254 τροπολογία Ντεμπάκερ που ζητά διαγραφή της σύστασης 6. Και αυτή την τροπολογία την ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για την παράγραφο 1 της ε, σύστασης 6 έχουμε την τροπολογία 255 Λόπε Φοντανία. ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 255 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας, 19 υπέρ, 20 κατά, μία απόχη, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την παράγραφο 5 της σύστασης 6 την τροπολογία 256 της κυρίας Λαπεφωτάνια υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 256 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας 23 ψήφοι υπέρ και 17 κατά εγκρίνεται 257 Λαπε Φοντάνια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 258 της ίδιας υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 259 της ίδιας υπέρ. Κατά. Ποιο είναι υπέρ επαναλαμβάνω. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σύσταση 7. Τροπολογία 260 του κ. Ντεπάκερ. Ζητά διαγραφή. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία μήμη υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 263. Ντεπάκερ ζητά διαγραφή τη σύσταση 8. Υπέρ, κατά, αποχέ Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 267 του κ. Ντεμπάκερ για τη σύσταση 9. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Σύσταση 10, 268 Φίλιπ Ντεμπάκερ. Και πάλι στα διαγραφή, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, οπότε ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία ομικρονόμικρον, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Γυρίζουμε λίγο πίσω και μετά τη συμβαστική τροπολογία νίνη θα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 264 της Ινέζου Μπέρ. Δεν είχε καταπέσει γιατί η 263 απορρίφθηκε. Προστίθεται μια νέα παράγραφος μετά την παράγραφο 8, λέει πρόεδρος. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 264 είναι Ζουμπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και παραρχόμαστε στην σύσταση 11 και τροπολογία 271 του κ. Ντεμπάκερ που ζητά διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία PP από δύο ομάδες. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Για την παράγραφο 3 της σύστασης 11 έχουμε την τροπολογία 272 της κυρίας Λόπε Φοντάνια που καταπίπτει. Οπότε περνάμε στη σύσταση 12 και την τροπολογία 273 του κυρίου Ντεμπάκερ που ζητά διαγραφή της σύστασης. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε την παράγραφο 1 της σύστασης 12 και την τροπολογία 274 Λόπε Φοντανία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, τι, τι είπατε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, ψηφίζουμε ολόκληρο το κείμενο ηλεκτρονικά. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 32 υπέρ, 5 κατά και 3 αποχές. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Et toute l'équipe de négociation. Le... Και όλη η διαπραγματευτική ομάδα. Το 21 αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη, οπότε περνάμε στο 22, όπου θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Δανούτα Γιαζοβιέτσκα που είναι γνωμοδότηση ουσιαστικά. Αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και θέμα τα εργαλεία για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Πρόκειται για την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Παριθμόν 25 του 2012. Παράγραφος 1. Συμβαστική D. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Τροπολογία 16 τη Αιγύτριας. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Η συμβαστική ε από 5 ομάδες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Συμβαστική F. 5 ομάδων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 6, τροπολογία 23 της εισηγητρίας, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6, τροπολογία 24 της εισηγητρίας με τροπορφορική τροπολογία της ιδίας. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, την ψηφίζουμε 24 υπέρ κατά. Αν δεν ψηφίζετε πια και απλώς ε, κουνιέστε, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Υπέρ λοιπόν κατά αποχές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Le vote est ouvert. Ψηφίζουμε. Pas pendant le vote. L'amendement est en vérification. Le vote est... Πέρασε τις ψηφοφορίες. 17 υπέρ, 18 κατά. Απορρίπτεται. Θέλετε να πάρετε το λόγο, κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που διαταράσω την ψηφοφορία, αλλά εξεπλάγει από την αρνητική στάση των σοσιαλιστών. Καταψήφισαν την τροπολογία που απλώς ζητά τα έγγραφα που λάβαμε για το 2014-2020 και τα σχετικά έγγραφα από το Κοινωνικό Ταμείο. Σε αυτά δεν μπορούμε να συζητούμε τώρα. Έχουμε ξεκινήσει την ψηφοφορία. Δεν έχετε δικαίωμα επέμβαση στο σημείο αυτό. Μετά την 24-25 του κυρίου Μπέκερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 του ιδίου υπέρ <clears throat> κατά αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονική για την 26. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Τέλος της ε, ψηφοφορίας, 31 υπέρ, 4 κατά, εγκρίνεται. 27 έχει αποσυρθεί, περνάμε στην παράγραφο 7, συμβαστική G. G, υπό 4 ομάδες, ε, υπέρ κατά αποχές, ε, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 7. Έχουμε την τροπολογία 31 του κυρίου Μπέκερ με προφορική της εισηγήτριας. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, στην προφορική τροπολογία ψηφίζω την, ψηφίζουμε 31. Όπως αποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές επαλήθευσης. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. 11 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας α, συμβαστική α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία, συμβαστική β, στο εκτιμώντας β, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από το εκτιμώντας β, τροπολογία 8, ριάμενρο, ήταν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9, της ιδείας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική σε από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το εκτιμώντας σε, τροπολογία 12, της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το ΣΕ, η τροπολογία 13 Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 33 pour, 2 contre, 0 abstention. Ε, Ωραία λοιπόν. Ε, εγκρίνεται ε, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και έτσι περνάμε στο σημείο 19. Et il s'agit du vote sur le rapport Πρόκειται για την ψηφοφορία επί της έκθεσης της συναδέλφου Μπάουερ για τα αποτελέσματα ε, των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για τα μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζόμενους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Έχουμε μόνο μία ψηφοφορία να κάνουμε που θα επικυρώσει τους καρπούς των διαπραγματεύσεων των οποίων ηγήθηκε η Edith Bauer και η διαπραγματευτική μας ομάδα. Θα ψηφίσουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 31 υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ε, Alors, attendez, attendez, attendez, ne partez pas tous. Ε, περιμένετε, ε, που πάτε, μην φύγετε όλοι. Έχουμε ένα σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι η ανταλλαγή με την ελληνική προεδρία. Είχαμε προβλέψει πως θα τελειώναμε τις ψηφοφορίες νωρίτερα, αλλά όχι και τόσο νωρίς. Οπότε η ελληνική προεδρία θα έρθει όπως λέει στα γαλλικά, ε, στο πικεφί. Θα έρθει λοιπόν στις 11 παρατέταρτο, γιατί τελειώσαμε πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαμε προβλέψει. Για το τεταρτάκι που έχουμε διάλειμμα και αν θέλετε να το διασκεδάσετε, δεν μπορώ να σας κλείσω την πόρτα, αλλά θα πρέπει να ξανάρθετε και έχουμε ακόμα δύο σημεία να εξετάσουμε. Οπότε σας ε, παρακαλώ να καθίσετε σιωπηλή. εδώ, στο σημείο 23. Ε... Prendre connaissance du projet d'avis σχέδιο γνωμοδότησης που σα παρουσιάζω εξ ονόματος της Επιτροπής μας ως συμβολή στην έκθεση πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει να συντάξει η Επιτροπή προπολογισμού με ε, γνωμοδότηση επί τη βάση του άρθρου 50 της Επιτροπής ΑΦΚΟ για τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της σύνταξης νομοδότησης λοιπόν, σας καλώ να διαπιστώσετε το εξής. Καταρχήν, και να τα σημειώσετε. Καταρχήν, ότι ο τρόπος με τον οποίο έγιναν αυτές οι διαπραγματεύσεις, κάνοντας διάκριση από τη μια πλευρά, ανάμεσα στην ε, διαπραγμάτευση για το νομοθετικό τμήμα και από την άλλη πλευρά του νούμερα, φάνηκε πως ήταν μια στρατηγική που αποδυνάμωσε την θέση του Κοινοβουλίου και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει ίσως αυτό να το σκεφτούμε. Δεύτερον, σας καλώ να σκεφτείτε αυτό που έγινε ότι δηλαδή χρειάστηκε να εργαστούμε επί των ε, αριθμών του 2011 που ήταν με αναθεωρημένα αλλά Σίγουρα δεν μπορέσαμε έτσι να λάβουμε υπόψη την εξέλιξη της κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος. Ε, σας καλώ ε, να δούμε σε ποιο βαθμό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έπαιξε πραγματικά το ρόλο του όταν πρόκειται για την νομοθετική διαδικασία. Και δεν θα αντισταθώ στο να σας ζητήσω να επανέλθετε εκ νέου στο θέμα του 25% και στον τρόπο με τον οποίο παρενέβη μια συνδεδεμένη επιτροπή στην Ολομέλεια όσον αφορά τις αποφάσεις που είχε λάβει μια άλλη επιτροπή. Επίσης σας καλώ να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας όσον αφορά τις συνθήκες εντό των οποίων χρειάστηκε να εργαστούμε, υπό τις οποίες μάλλον χρειάστηκε να εργαστούμε για την έκθεση Χάρκιν για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, αυτό της κυρίας Κοστέλο που αφορούσε το ε, Ταμείο για τους, πιο, για τους απόρους. Ε, ε, πράγμα που δεν μας επέτρεψε να πάμε μέχρι εκεί που θα επιθυμούσαμε, αν και τελικά ικανοποιητικό είναι το αποτέλεσμα. Ε, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο διοργάνωσε τις διαπραγματεύσεις το Κοινοβούλιο για τη διαπραγμάτευση των οριζόντιων προγραμμάτων θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Επίσης πιστεύω ότι Ο τρόπος με τον οποίο προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις για τις νομοθετικές βάσεις στο πλαίσιο το γενικότερο των διαπραγματεύσεων δημιούργησε πρόβλημα και προτείνουμε τέλος να σκεφτούμε την, το ενδεχόμενο το Συμβούλιο, διαχειριζόμενο τη σχέση με το Κοινοβούλιο επί τη βάση μερικής προσέγγισης ή γενικής προσέγγισης, ε, ε, να μην ε, σεβάστηκε απόλυτα το πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Σε αυτό το στάδιο αυτά έχω να σας πω και μπορώ να σας πω ήδη ότι χρειάζεται να ενεργήσουμε για διάφορα στοιχεία και να παρέμβουμε για τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωκοινοβούλιο βελτίωσε την προπαρασκευαστική εργασία που είχε κάνει στο πλαίσιο της, της Επιτροπής ΣΟΥΡ ε, θα λάβουμε βεβαίως υπόψη τις παρατηρήσεις της ίδιας της Κομισιόν επ' αυτού, αλλά έχω την εντύπωση πως ίσως θα μπορούσαμε εδώ να προχωρήσουμε περισσότερο. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει μια ολόκληρη σειρά τροπολογιών, αλλά με τα χαρά θα δεχτώ και τις συμβολές των μελών όσον αφορά διαδικαστικά θέματα και κυρίως το, ένα θέμα πολύ σημαντικό όπως αυτές οι νομοθετικές βάσεις στο πλαίσιο των πολιετές όπου στην ουσία, ή μάλλον η Κομισιόν μας έπνιξε με ένα σωρό νομοθετικές προτάσεις, πράγμα που όσον αφορά τον ορισμό των στρατηγικών και των πολιτικών προτεραιοτήτων δεν μας δίνει την καλύτερη ορατότητα. Και από την άποψη ε, της διαδικασίας δεν βρίσκω φυσιολογικό σε, για μικρές νομοθετικές βάσεις να πάμε με διαπραγματευτικές εντολές ε, πολύ μαχητικές και εδώ που στην ουσία η Κομισιόν είχε, να ασχοληθεί με το θέμα του κοινωνικού ταμείου να μπει στη διαπραγματεύση χωρίς έντολη από την Ολομέλεια. Και τέλος να ξαναπώ και να αναφέρω τα ραντεβού που έχουμε και στα οποία δίνουμε μεγάλη σημασία στην υιοθέτηση της νομικής βάσης στο ραντεβού που δώσαμε με τους συνομοθέτες για το μέλλον της εγγύησης για την νεότητα. Αυτά είχα να πω και όποιος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο. Σα ε, κυρία Χάρκιν και μετά η Τζιν Λάμπερτ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για το σχέδιο χνομοδότησης που συντάξατε Σύμφωνο με όλα όσα είπατε, εγώ δεν συμμετείχα, είχα όμως συμμετοχή στο ETF και γνώριζα τι συμβαίνει. Νομίζω πως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα σε αυτή τη διαδικασία απόφασης είναι σημαντικό και πρέπει όλα αυτά να τα εκμεριωθούν γιατί θα έχουμε νέο κοινοβούλιο και κάποιοι δεν θα έχουν την εμπειρία που αποκομίσαμε εμείς αυτή τη φορά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταγραφούν τα διδάγματα που αποκομίσαμε και να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Για το Συμβούλιο βεβαίως ήταν κάτι το πολύ νέο και το, θέμα της ε, εξουσίας και της επιρροής που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Για την παράγραφο 2 εδώ δεν είμαι απόλυτα βέβαιη το τι εννοεί. Λέει λυπάται που η, τα, τα νούμερα του 2011 που προτέθηκαν από την Κομισιόν ως βάση για τις διαπραγματεύσεις δεν αντικατόπτυζαν την πραγματικότητα των κρατών μελών. Ε, εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα πρόβλημα διατύπωσης εδώ. Για το κοινωνικό ταμείο και για το Σαπόρους υπήρχε χρονική πίεση, αλλά και για άλλα πράγματα υπήρχε χρονική πίεση και επίσης συμφωνώ πως η διαίρεση των διαπραγματεύσεων σε νομοθετική βάση και σε νούμερα μας αποδυνάμωσε. Γιατί ενώ προσπαθούσαμε να πετύχουμε το ένα, χάναμε το άλλο. Και ήταν πολύ δύσκολο να τα συνδυάσουμε όλα μαζί. Αλλά όπως είπα, θα, εγώ έχω συζητήσει γι' αυτό πολύ με τους συναδέλφους και ελπίζω πως θα μπορέσω να συντάξω κάποιες τροπολογίες για το κείμενο. Ευχαριστώ Γιτζίνε Λάμπερτ. Ευχαριστώ και εγώ. Συμφωνώ ο γενικός και τα όσα είναι εδώ καταγεγραμμένα και στηρίζω και τη Μάριον Χάρκινγκ στα όσα μόλις είπε. Ε, νομίζω πως υπάρχει επίσης θέμα για ε, σε εσωτερικές ε, ανακοινώσει μάλλον του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη μετακίνηση των διαπραγματευτικών θέσεων που που δεν ε, ανακοινώνονταν πάντα, δεν υπήρχε επικοινωνία εν πάση περιπτώσει και δεν συζητώνταν πάντα οι αλλαγέ. Δηλαδή, πιστεύαμε πως κάποια πράγματα θα συζητώνταν, αλλά δεν συζητώνταν πλέον λόγω αποφάσεων που είχαν ληφθεί αλλού. η έλλειψη διαπραγματευτικής πίεσης από την Ολομέλεια δεν μας βοήθησε στο να πετύχουμε ε, το αποτέλεσμα που θέλαμε από πλευράς Κοινοβουλίου. Θα το δούμε λοιπόν στην ομάδα μας, θα συνομιλήσω με όσους συμμετείχαν πιο άμεσα. Εγώ τα κατάφερα και έβγαλα την ουρίτσα μου απ' έξω σε όλη τη διαδικασία, αλλά θα επανέλθω. Πάντως συμφωνούμε με τις επικρίσεις και με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και χαίρομαι που τα μέλη της Επιτροπής μας ε, ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτή την αξιολόγηση και είναι αυτό που ε, κίνησε το γενικό ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε ακριβή και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, τεκμηριωμένη αξιολόγηση για το σύνολο της διαδικασίας. Με ιδιαίτερη έμφαση στην πτυχή απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις. Συμφωνώ με την κυρία Χάρκιν ότι στην παράγραφο 2 θα πρέπει να πούμε στα κράτη-μέλη. Βέβαια είναι κάπως συμβιλικό το κείμενο και χρήζει τροποποίησης, αλλά για το 2011 αυτό που λείπει είναι σε σταθερές τιμές. Αυτή η φράση. Γιατί, αν δεν κάνω αυτό έλεγε και το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2011 σε σταθερές τιμές. Αυτό όμω δεν αλλάζει τίποτα, γιατί στην Ιρλανδία έχουν αλλάξει τα πράγματα άρδιν. Και όταν συζητούσαμε την εγγύηση για του νέου το Youth Guarantee, το θέμα των ποσών και των αριθμών για το 2012 δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα της Ιρλανδίας. Και γι' αυτό τροπολογήσαμε την παράγραφο. Έχουμε και μία προθεσμία για τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης που λήγει στις 28 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες μόνο στα αγγλικά τροπολογίες. Οι συμβαστικέ τροπολογίε θα εξεταστούν στις 12 Φεβρουαρίου, θα ψηφίσουμε στις 13. Η Επιτροπή Προπολογισμών θα ψηφίσει 6 Μαρτίου και θα πάει το θέμα στη Ρολομέρεια του Απριλίου. Πρώτο τελευταίο θέμα της σα διάταξη. το 24, ο κύριος Νταρντέν θα μα ενημερώσει για τη διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο σχετικά με τη ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόληση ε, που έγινε χθε. Ο κύριος Νταρντέν. Ευχαριστώ. Όντω, χθε έγινε η δεύτερη συνάντηση του τριμερούς διαλόγου με θέμα της δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Στην αρχή η ελληνική προεδρία μας είπε ότι είχε ελάχιστο περιθώριο λιγμών μετά την πρώτη ενημέρωση που έγινε στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, την Κορεπέρ, αλλά η ελληνική προεδρία είχε βούληση και επιθυμία να διεκπαιρεώσουμε το θέμα και θα επιδείξει δημιουργικό και συνεργάσιμο πνεύμα. Αυτό χρειαζόμαστε και από τις δύο πλευρές, ευρηματικότητα και δημιουργικότητα. Για ορισμένα σημεία είχαμε ικανοποιητική συμφωνία. Για παράδειγμα, έχουμε τον ορισμό του bench learning. Επίσης, έχουμε μία παρουσία στοιχείων σε, και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που χρειάζεται και σε περίπτωση που έχουμε περιφερειακή οργάνωση για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης θα συμπεριληφθούν αυτές τις δραστηριότητές μας. Αλλά και για τη νομική βάση καταλήξαμε σε ικανοποιητική συμφωνία επιμένοντας τον ε, δωρεάν χαρακτήρα που θα πρέπει να έχουν αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Τρία σημαντικά θέματα συζητήθηκαν χθε στις διαπραγματεύσεις. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης στο δίκτυο, εμείς ε, εμείναμε στην πρότασή μας για προαιρετικό χαρακτήρα, γιατί θα ήταν πρόωρο να πούμε τελικά ότι συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο, αλλά καταθέσαμε συμβαστική πρόταση που ζητά επαναφορά στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ουσιαστικά υπαναχωρήσαμε σε σχέση με μερικές τροπολογίες μας στην Επιτροπή, αλλά ζητήσαμε και από το Συμβούλιο να αποσύρει κάποια σημεία που είχε εντάξει το κείμενο, επιμένοντας ε, εμείς στον προαιρετικό χαρακτήρα και συντάξαμε μια τελογική σκέψη που επέμεινε στην παρουσία αυτών των υπηρεσιών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά προτείναμε στο Συμβούλιο και ελπίζω να τα δεχτεί η Κορεπέρ. Σε ό,τι αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης, ένα άλλο σημαντικό θέμα, και εκεί υποβάλαμε συμβαστική τροπολογία που λέει είτε να μπουν στο κείμενο της απόφασης, στο διατακτικό της απόφασης, στους άξονες δραστηριοτήτων, στις πρωτοβουλίες, στο bench learning, bench learning, learning. Ε, και είπαμε ε, ίσως μπουν οι δείκτες στο παράρτημα και περιμένουμε την πρόταση για τους δείκτες, τους ποιοτικούς και τους ποσοτικούς και επίσης για το Διευθυντήριο προβλέπονται κάποιες εξουσίες που θα πρέπει να διευκρινιστούν εσωτερικά. Μέχρι στιγμής από τις διαπραγματεύσεις προέκυψε ότι οι δείκτες θα μπορούμε κατά εξουσιοδότηση πράξης να αναθεωρούνται και να συμπληρώνονται, αλλά οι κατεξουδότηση πράξη θα περιορίζονται σε αυτό μόνο το θέμα. Αυτά για το δεύτερο θέμα. Τώρα για το τρίτο θέμα των διαπραγματεύσεων. Την παρουσία δηλαδή στο δίκτυο του ΕΜΚΟ για τη βελτίωση της συνεργασίας ε, και της ε, σωστής ε, διάδοσης των πληροφοριών, διαβίβαση των πληροφοριών. Εμείς συζητήσαμε το ΕΜΚΟ να έχει καθεστώς παρατηρητή και να μην είναι συστηματικός ο χαρακτήρας παρουσίας του θα συγκεκριμενοποιηθεί η συμβαστική τροπολογία ε, και θα λέμε ότι η ΕΜΚΟ δεν είναι στο δίκτυο αλλά στο διευθυντήριο εκτός και αν γίνονται περιορισμένες ε, συνεδριάσεις. Τώρα τι είδους ε, συνεδριάσει κλειστό κύκλο ή και κλεισμένο το θηρό. Θα δούμε, θα διευκρινιστεί αυτό στην επόμενη μας πρόταση, ώστε να μπορέσει η Προεδρία να καταθέσει το κείμενο στην Κορεπέρ. Τώρα, τι με έλεγε Νέστε. Την επόμενη Τετάρτη προβλέπεται νέο τριμερή διάλογο που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και ο τελευταίο. Θα έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών και προτάσεις και αντιπροτάσεις για τη διατύπωση και ίσως μια-δυο τεχνικές συνεδριάσεις για να επιλύσουμε τις εκκρεμότητες. Αυτά κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ακριβή αυτή παράθεση των τεχθέντων. Σημασία για την παρουσία της ΕΜΚΟ από, για το Συμβούλιο είναι σημαντική. Χωρίς ωστόσο την κατεύθυνση της ΕΜΚΟ και από την άλλη μεριά για τον υποχρεωτικό ή μη χαρακτήρα του δικτύου. Η απόφαση του Συμβουλίου είναι απολύτως ακατανόητη. Μία ερώτηση πρέπει να θέσουμε στο Συμβούλιο. Εάν υπάρχει ειδική πλειοψηφία υπέρ του προερωτικού χαρακτήρα. Γιατί αρχίζω και έχω αμφιβολίες σε σχέση με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ερμηνείας που δίνεται στον τριμερή διάλογο γιατί το δίκτυο είναι υποχρεωτικό. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο επιθυμεί τώρα να ανοίξει το θέμα του ενδεχόμενα προαιρετικού χαρακτήρα ξυλώνει σε μεγάλο βαθμό ακόμα και τον λόγο ύπαρξης διαδικασίας. Και το Κοινοβούλιο έχει δίκιο να το σημειώσει και να επιμείνει ώστε οι δέσμοι όπως προτάθηκε στο Συμβούλιο μετά από τη δική σας πρόταση χθε, ότι για μας είναι απαράβατο όριο, είναι κόκκινη γραμμή δηλαδή, που δεν μπορεί να τη διαβεί κανείς. Ολοκληρώσαμε τώρα το θέμα αυτό. Υπάρχουν άλλες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ε, κυρία ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση του θέματος για τις συζητήσεις που έγιναν τώρα για τους δείκτες. Γνωρίζω ότι είναι σημαντικό διότι το ποσοστό της ανεργίας και της απασχόλησης υπάρχουν δείκτες οι οποίοι απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο ή εξαντιθέτου... όχι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στις διαπραγματεύσεις για τους δείκτες αναμένουμε την πρόταση που θα κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μεσημέρι και μόλις θα έχουμε την πρόταση αυτή θα εξετάσουμε προσεκτικά το θέμα αυτό και θα αντιδράσουμε μέχρι το βράδυ στις 8 για να μπορέσει το Συμβούλιο μετά να προχωρήσει στην ε, μόνιμη αντιπροσωπεία Κορεπέρ την Παρασκευή. Θα μας εξηγήσει μετά ο εισηγητής μας το τι θα γίνει στον επόμενο τριμερή διάλογο που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου όπως εξήγησε ο ίδιος και θα τα πούμε στο Στρασβούργο. Σας παρακαλώ λοιπόν να μείνετε διότι πρόκειται να προσέλθει ο Έλλην Υπουργός.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 Euh, Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις ενημέρωσα τον κύριο Υπουργό για την συζήτηση που διεξαγάγαμε για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχολήσεως, διότι είναι ένα θέμα το οποίο τον απασχολεί και τον ίδιο και μας άλλωστε και γνωρίζουμε πόσο η ελληνική Προεδρία κινητοποιείται για να προωθήσει ολόκληρη αυτή την νομοθετική συζήτηση και τις άλλες συζητήσεις που βρίσκονται ακόμα επιτάπητος και όχι μόνο διότι υπό την Προεδρία σας που για μας θα είναι και η τελευταία, στην ε, παρούσα κοινοβουλευτική θητεία δηλαδή, μένουν ακόμη πολλά πράγματα ανοιχτά, πολλά θέματα ανοιχτά, από την σκοπιά νομίζω το, της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Vous avez... Euh, Έχετε λοιπόν εσείς τις δικές σας προτεραιότητες, εμείς έχουμε τις δικές μας είναι, έχει έλθει η ώρα να ανταλλάξουμε προτεραιότητες για να εξασφαλίσουμε ώστε αυτή η τελευταία προεδρία στη διάρκεια της της κοινοβουλευτικής θητείας να είναι και η αυτή που θα δείξει τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ προεδρίας και Επιτροπής Απασχολήσεως και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήδη είδαμε την δέσμευσή σας διότι είδαμε και στην Αθήνα σε διαφορετικές ε, συνθέσεις, σας έχουμε δει δηλαδή, σας είδαμε και από την αρχή της εβδομάδας, αν μπορώ να το πω έτσι, εδώ στις Βρυξέλλες και την δέσμευση σας για το πολύ σημαντικό θέμα των σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και των σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια για θέματα προϋπολογισμών και την διαπραγμάτευση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σήμερα βεβαίω είστε παρόν εδώ για να παρουσιάσετε τις δικές σας προτεραιότητε, και θα σα δώσω ευχαριστώ το λόγο για να το πράξετε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, ενώπιον των εκπροσώπων των πολιτών της Ευρώπης. Το Ευρωκοινοβούλιο συνιστά βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, γιατί μεταφέρει αυθεντικά τον παλμό, τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις ελπίδες των Ευρωπαίων πολιτών. Και κάτι ακόμα. Οι ευρωβουλευτές στην πλειοψηφία τους όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο στάθηκαν δίπλα στην Ελλάδα. Κάτι που ο ελληνικός λαός δεν θα ξεχάσει ποτέ. Σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Ιστορικά τις μεγαλύτερες, θα έλεγε κάποιος, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκλήσεις που όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά. Η Ελλάδα βίωσε εντονότερα από κάθε άλλο κράτο μέλος τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Η κρίση στη χώρα μου δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο των εσωτερικών διαρθρωτικών αδυναμιών της, αλλά αποτέλεσμα και των δομικών αδυναμιών του ίδιου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία σε μια συγκυρία που απαιτεί τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Αποφάσεις για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Αποφάσεις για την πρόθεση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Αποφάσεις για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αποφάσεις που θα αποτελέσουν απάντηση και θα αποκλείσουν τις ακραίες αντιευρωπαϊκές φωνές λαϊκισμού που εκμεταλλεύονται την κρίση για να ακουστούν αλλά και να μειώσουμε την επιρροή όσων δεν θέλουν την Ευρώπη ενωμένη. Αποφάσεις αναγκαίες που πρέπει να πάρουμε τώρα, ώστε στις επικείμενες ευρωεκλογές που συμπίπτουν με το τέλος της ελληνικής προεδρίας, οι Ευρωπαίοι πολίτες να μην ψηφίσουν με την πικρή γεύση της κρίσης. Τώρα δύο λόγια για την Ελλάδα που με το ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που συνεχίζει να υλοποιεί αλλά και τις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού εμφανίζει τις πρώτες θετικές ενδείξεις. Συγκεκριμένα, η ανεργία το 2013 σταθεροποιήθηκε, ενώ για το 2014 αναμένεται για πρώτη φορά η σταδιακή αποκλιμάκωσή της. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα παρουσιάσει για πρώτη φορά πλεόνασμα το 2013 μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα θα εμφανίσει επίσης για πρώτη φορά πρωτογενές πλεόνασμα μετά από 10 χρόνια. Στόχο που πετυχαίνουμε μάλιστα ένα χρόνο νωρίτερα από τις προβλέψεις του προγράμματος. Το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά που η οικονομία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη μετά από έξι χρόνια ύφεσης. Και τέλος, ο ίδιος ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης συμπεριέλαβε την Ελλάδα ως πρώτη χώρα σε μεταρρυθμίσεις. Αξιότιμη μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήδη διανύουμε το πέμπτο έτος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων αυτής στρατηγικής, η Ελληνική Προεδρία έχει διαρθρώσει τις προτεραιότητές της στο πεδίο της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, πάνω σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτος άξονας. Η πρόθεση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας. Δεύτερος άξονας. Η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ. Τρίτος άξονας η πρόθεση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα. Η ελληνική προεδρία θα κινηθεί με αποφασιστικότητα επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξής κατευθύνσεις. Πρόθεση της ουσιαστικής ένταξης της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου περαιτέρω βελτίωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση του πίνακα αποτελεσμάτων scoreboard που αποτελεί σημαντική κατάκτηση για την κοινωνική Ευρώπη. Ήδη έχουν υποβληθεί ουσιαστικές προτάσεις για την ενίσχυση του πίνακα με νέους κοινωνικούς δείκτες. Από τη δική μας πλευρά και λόγω του γεγονότος ότι η Ευρώπη γερνάει θα βλέπαμε αναγκαία την ενσωμάτωση της δημογραφικής διάστασης στον πίνακα των αποτελεσμάτων. Ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ σημαίνει διάλογος, συνένεση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες της Ένωσης. Η τρέχουσα κοινωνική και εργασιακή κατάσταση απαιτεί σήμερα περισσότερο από ποτέ τη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Η Ελληνική Προεδρία θα εργαστεί για την υιοθέτηση της απόφασης που ενισχύει τη θεσμική διάσταση της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής. Για το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων, posting of workers. Το Συμβούλιο Απασχόλησης ΕΠΣΚΟ στις 9 Δεκεμβρίου έλαβε μια πολύ σημαντική και συμβολική απόφαση. Η απόφαση αυτή είναι η απόδειξη της πολιτικής βούλησης των κρατών μελών και σας διαβεβαιώ ότι η ελληνική προεδρία θα αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία προκειμένου η διαδικασία τριλόγου που έχει ξεκινήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καρποφορήσει. Γνωρίζω τις δυσκολίες. Ωστόσο, ανοίξαμε μία πόρτα και δεν πρέπει να την κλείσουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα της αποτυχίας. Το εγχείρημα είναι δύσκολο, καθώς θα πρέπει να συγκεραστούν διαφορετικές απόψεις. Αυτή όμως είναι η δύναμη της Ευρώπης. Ο συγκερασμός των απόψεων. Το μέλλον της Ευρώπης είναι οι νέοι της Ευρώπης. Γι' αυτό θα δώσουμε τη μάχη με ό,τι όπλα διαθέτουμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το νοσηρό φαινόμενο της ανεργίας των νέων. Γι' αυτό η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητές μας. Στόχος μας είναι να παρακολουθήσουμε από κοντά την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος «Εγγύηση για την νεολαία» Youth καρατί, και να εμβαθύνουμε τις πρωτοβουλίες σε αυτό το τομέα. Επιπλέον με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για την ομαλή μετάβαση των νέων στον εργασιακό βίο θα προωθήσουμε την υιοθέτηση μιας σύστασης που θα θέσει το ποιοτικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση. Έτσι, θα διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν υψηλής ποιότητας προγράμματα πρακτικής άσκησης, γεγονός ύψης της σημασίας στον αγώνα κατά της ανεργίας των νέων. Επίσης, στις προτεραιότητές μας είναι η πρόθεση της συνεργασίας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση στις 9 Δεκεμβρίου σχετικά με την απόφαση για τη βελτίωση αυτής της συνεργασίας. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά μια ευρεία συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό τη θεσμική κατοχήρωση του δικτύου. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της διαδικασίας τριλόγου μας δίνουν βάσιμα τη δυνατότητα να πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Η βελτίωση της κινητικότητας και η επίτευξη συμφωνίας για μια γενική προσέγγιση για τον κανονισμό επανασύστασης του Γιούρες αποτελεί άλλο ένα στόχο της ελληνικής προεδρίας. Το Συμβούλιο χαιρετίζει τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Καθώς θεωρεί ότι το αναθεωρημένο Γιούρες αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα εργαστούμε με μεθοδικότητα για την καταπολέμηση του απαράδεκτου φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, του οποίου τις αρνητικές επιπτώσεις αναγνωρίζουμε όλοι. Η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας απαιτεί τήρηση νομιμότητας. Εμείς ως χώρα, δυστυχώς μέχρι πρόσφατα, είχαμε πολύ υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας. Προσωπικά την αδήλωτη εργασία την έχω χαρακτηρίσει ως οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα στερεί σημαντικούς πόρους από το ασφαλιστικό σύστημα, υπονομεύει τον υγιή ανταγωνισμό και τις συνεπείς επιχειρήσεις και το χειρότερο παραβιάζει τα εργασιακά δικαιώματα. Πρόσφατα στην Ελλάδα, για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού, προχωρήσαμε στη λήψη δέσμης μέτρων με την κωδική ονομασία Άρτεμις. Και σήμερα τέσσερις μήνες μετά την πρώτη εφαρμογή τους, είδαμε ότι τα μέτρα έπιασαν τόπο. Χτυπήσαμε το κακό στη ρίζα του. Πιστεύουμε ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μολονότι υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στο συγκεκριμένο τομέα, εν είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε μια κοινή απόφαση για τη δημιουργία πλατφόρμας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Επιπλέον, εντός των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας συμπεριλαμβάνεται το ζήτημα των ίσων ευκαιριών και της μάχης κατά των διακρίσεων. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, η ελληνική προεδρία θα εξετάσει την πρόταση για μια οδηγία για την ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την πίστη, την αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό. Επιπλέον, θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση της υιοθέτηση της πρότασης για μια οδηγία για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Κυρίες και κύριοι, σήμερα περισσότερο από ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από δημοσιονομική σταθερότητα, και εμβάθυνση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η κοινωνική συνοχή αποτελεί ταυτόχρονα προαπαιτούμενο αλλά και συνέπεια της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Για να ξεπεράσουμε την κρίση, για να αναδυθούμε την επόμενη μέρα της κρίσης, ως Ένωση δυνατότερη πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην κοινωνική Ευρώπη. Το πρόγραμμά μας είναι φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικό. Εγώ προσωπικά από το βήμα αυτό αλλά και όλοι οι συνεργάτες μου θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα εργαστούμε με επιμονή, υπομονή και αποφασιστικότητα για μια πετυχημένη ελληνική προεδρία. Γιατί επιτυχημένη ελληνική προεδρία σημαίνει επιτυχία και της ίδιας της Ευρώπης επιδιώκω τη στενή συνεργασία μαζί σας. Γιατί μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αν διασταυρώσουμε τα ξύφη των ιδεών μας, θα πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους και τα κοινά μας οράματα. Είναι υποχρέωση και καθήκον μας, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις επόμενες γενιές της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τα πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί. Επιθυμεί άλλος κανείς. Η κυρία Εσαγιά. Κυρία Μανικατού. Ωραία, κλείνω λοιπόν εδώ τον κατάλογο των εγγεγραμμένων. Ο κύριος Σέρκας πρώτος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ και εσείς και το επιτελείο σας. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην Επιτροπή μας και σας ε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην Αθήνα και για την αγαστή συνεργασία που έχουμε ιδιαίτερα για την έκθεσή μου, για τη συνέπεια των προγραμμάτων της Τρόικας στις τρεις χώρες που εφάρμοσαν το μνημόνιο. Ευελπιστώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η αγαστή συνεργασία, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να αναφερθώ στα πρώτα σας λόγια. Πιστεύω ότι όντως η Ελλάδα έχει τεράστιες προκλήσεις να αντιμετωπίσει εσωτερικές, αλλά και μεγάλες προκλήσεις ε, κατά την άσκηση της Προεδρίας σας. Πιστεύω ακράδαντα όμως ότι θα στεφτεί με τεράστια επιτυχία η ελληνική Προεδρία και θα είναι επιτυχία και θρίαμβος και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Γιατί πιστεύω ότι παρά τη συγκυρία και παρά τις ε, μεταβαλλόμενες απόψεις, όταν δει κανείς σε βάθος τα πράγματα, διαπιστώνει ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να φανταστεί την Ελλάδα εκτός της Ευρώπης. Και κανένα ε, λογικό άνθρωπο που έχει σώσει τα σφρένα δεν θα μπορούσε να φανταστεί την Ευρώπη χωρί Ελλάδα. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα κτίριο χωρί τα θεμέλια του. Έτσι θα ήταν αν φανταζόμασταν την Ευρώπη χωρί έναν ακρογωνιαίο λίθο όπω τη Ελλάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα αξιοποιήσουν αυτό το εξάμεινο για να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες αυτές προκλήσεις. Και χαίρομαι που έχετε καλά μακροοικονομικά στοιχεία. Και ευελπιστώ ότι ο ελληνικός πληθυσμός που τόσο έχει υποφέρει, τόσο έχει ταλανιστεί ε, και τόσο έχει υποστεί επιθέσεις και ταπεινώσεις και εξευτελισμούς να, να αποκτήσει την αισιοδοξία με αυτά τα καινούργια στοιχεία. Εμείς ανέκαθεν ε, είχαμε εμπιστοσύνη και είχαμε μεγάλη κατανόηση προς την Ελλάδα και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι η πικρή γεύση της κρίσης ίσως θα πρέπει κάπως να μετριαστεί από τις πολιτικές για την κρίση. Γιατί οι πολίτες της Ελλάδας αλλά και ε, της Νότιας Ευρώπης ε, σε αυτή την πικρή γεύση της κρίσης δυστυχώς έχουν να προσθέσουν και την πικρή γεύση από τις πολιτικές που εφαρμόσαμε για την κρίση. Δυστυχώς δεν ήταν θετικές. Ήταν αναποτελεσματικές αυτές οι πολιτικές και άδικες. Και μπορεί ο κόσμος να είναι έτοιμος να κάνει θυσίες και να αντιμετωπίσει προκλήσεις, αλλά αν αυτές οι προκλήσεις και τα μέτρα είναι δίκαια και αναλογικά και όχι αδυσόπιτα και δρακόντια. Γιατί ε, περίμεναν μία επέμβαση από χειρούργους ε, οι λαοί μας και τελικά βρέθηκαν απέναντι σε χασάπιδες που κρατούσαν ε, ε, Δρεπάνη και χασαπομάχαιρο. Τέτοια ήταν τα μέτρα τα δρακόντια. Μιλήσατε για το posting, την απόσπαση εργαζομένων και τις άλλες δύο οδηγίες ε, ε, για τις μετακινήσεις εσωτερικά στις επιχειρήσεις και τους εποχικούς εργαζομένους. Ελπίζω να δείξετε συνεργάσιμο, συνεργάσιμο πνεύμα και να μετακινηθεί κάπως η θέση του Συμβουλίου. Γιατί φαίνεται ότι για το Συμβούλιο διάλογο σημαίνει πλήρη αποδοχή της θέσης του Συμβουλίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι, δεν είναι αυτός ο διάλογος. Ελπίζω λοιπόν να συνεχιστεί πραγματικός διάλογος και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Προεδρία. Ας, ακούσουμε ακόμη δύο. Τζιν Λάμπερτ και μετά θα ακολουθήσει ο κ. Πουπάκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την νέα Προεδρία για την ανάπτυξη των προτεραιοτήτων της. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη και εγώ και η πολιτική μου ομάδα την έμφαση που δίνεται στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης στη διαδικασία του εξαμήνου. Καλή τύχη, σας ευχόμαστε. Είναι κάτι το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το προωθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζουμε όμως ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτιώσεων. Χαίρομαι επίσης για τα όσα είπατε για τον κοινωνικό διάλογο. Ερώτηση για τον διάλογο της κοινωνίας των πολιτών επίσης, που είναι κάτι το οποίο λείπει κατά τη γνώμη μας σε πολλές χώρες μέλη στη διαδικασία του εξαμήνου. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω εάν ο διάλογος της κοινωνίας των πολιτών επίσης ή με την κοινωνία των πολιτών επίσης θα αποτελέσει μέρος της ατζέντα σας. Και σε ό,τι αφορά την αδήλωτη εργασία, γνωρίζω ότι αυτό υπήρξε προτεραιότητα και προηγουμένων προεδριών, δεν ξέρω με πόση επιτυχία την πρόθεσαν. θα ήθελαν να ρωτήσω με ποιο τρόπο θα προσεγγίσετε το θέμα σε σχέση με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας. Διότι συμφωνούμε μεν ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι που έχουν δουλειά να είναι και ενταγμένοι στα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας, γνωρίζουμε ωστόσο ότι ορισμένα συστήματα δεν ανταποκρίνονται και ιδίως όταν ορισμένοι έχουν πολύ σύντομε σύντομου χρόνου συμβάσει εργασία ή άτυπε συμβάσει εργασία και μπαίνουν και βγαίνουν στα συστήματα αυτά κοινωνική ασφάλεια, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο Ενωμένο Βασίλειο έχουμε πολλού που χρησιμοποιούν τι τράπεζε τροφίμων. Αναγκάζονται να καταφεύγουν σε αυτέ, διότι τα συστήματα κοινωνική ασφάλεια δεν του προλαβαίνουν όταν αυτοί μπαίνουν, βγαίνουν στα συστήματα, διότι έχουν πάρα πολύ ε, πρόσκαιρε συμβάσει εργασία. Ποια θα είναι η προσέγγιση σας λοιπόν θα δεν είναι μονάχα η κατασταλτική πλευρά. η τη εργασία, η επιβολή ποινών κτλ. Πρέπει να δείτε και την άλλη πλευρά, να μπορέσετε να βοηθήσετε να γίνουν οι αλλαγέ που είναι απαραίτητε. Κύριε Πουπάκη, εσεί τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια κύριε Υπουργέ ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε μια περίοδο που η ενίσχυση τη κοινωνική διάσταση στην ΟΝΕ βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διεργασιών και κυρίως αποτελεί πλέον αναγκαία συνθήκη διαβίωσης για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο ότι η χώρα που καλείται να θεμελιώσει την απαιτούμενη ισορροπία, τη συμφιλίωση δηλαδή μεταξύ δημοσιονομικής εξυγίασης και κοινωνικής συνογής, είναι η χώρα που η κοινωνία της έχει υποβληθεί στις πλέον δυσβάστακτες θυσίες, χάνοντας το 50% του βιωτικού του επίπεδου, με την ανεργία του 27%, με την αγοραστική δύναμη των μισθωτών να μειώνεται κατά 37% την τελευταία τετραετία, Περίπου ένα στα πέντε νοικοκυριά αναγκάζονται να ζήσουν χωρί εισόδημα, η φτώχεια να αυξάνεται δραματικά και στι πιο ακραίε τη μορφέ κλπ. Έχοντα λοιπόν σαν δεδομένο ότι τα ωφέλη τη ανάπτυξη επιβάλλεται να διαχέονται σε όλο το φάσμα του κοινωνικού ιστού, αλλά και ότι όσο διευρύνονται οι εισοδηματικέ ανισότητε και το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών μεγαλώνει, τόσο μεγαλύτερα, θα, περισσότερο θα απειλείται η κοινωνική αλλά και η οικονομική σταθερότητα. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή μιλήσατε για του δείχτε να ρωτήσω πώς σχεδιάζει η ελληνική Προεδρία να προωθήσει στην πράξη το ζήτημα της ενσωμάτωσης των κοινωνικών δικτών στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά και προτίθεται η ελληνική Προεδρία να αναλάβει πρωτοβουλίες για την έκδοση ειδικών αναχώρα συστάσεων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ελλημάτων στα κράτη-μέλη που βρίσκονται υπό το καθεστώς των μνημονίων. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας προτείνω να απαντήσετε σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Έχουμε ακόμα πέντε ερωτήσεις, ε, παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Ξεκινάω από τον Αλεξάνδρο Σέρκας, με τον οποίο πρέπει να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση μέσα από την ανταλλαγή απόψεων όλο αυτό το διάστημα, σχέση η οποία συνεχίστηκε και με την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα και εκ προημίου θέλω να πω για συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνατε όσο αφορά το κείμενο για τις επιπτώσεις που είχε στην Ελλάδα όλη αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή. Ένα κείμενο που στον πυρήνα του δείχνει και το χαρακτήρα σας, ότι είσαι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία με την Τρόικα, μια σκληρή διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε ένα ευρύ πλαίσιο μεταρρυθμίσεων και απομένει κι άλλο ένα τμήμα, πολύ λίγο πλέον, δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης όσο αφορά το θέμα της Τρόικα και τη συνεργασία μαζί της είναι ήδη αναρτημένες στο ίντερνετ διαμέσου του Υπουργού Οικονομικών του κ. Στουνάρα και είναι στη διάθεση όλων. Από εκεί και πέρα απομένουν όπως είπα λίγα ακόμα για την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τα οποία η ελληνική κυβέρνηση θα τα προχωρήσει. Ε, υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την άλλη πλευρά. Οι μεν δείκτες, οι δημοσιονομικοί δείχνουν για πρώτη φορά σας τους περιέγραψα πρωτογενές πλεόνασμα, αρχίζει να αποκλιμακώνεται η ενεργία το 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα είναι θετικό για πρώτη φορά, περνάμε σε ανάκαμψη από ύφεση 6 ετών, όλα αυτά είναι τα θετικά. Δυστυχώς όμως το αποτύπωμα της κρίσης και αυτής της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής άφησε πίσω της έντονα κοινωνικά αχνάρια, αποτυπώματα. Δηλαδή η ανεργία στην Ελλάδα σήμερα έχει εκτιναχθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ύψος, δυστυχώς το υψηλότερο στην Ευρώπη και το πιο δυσάρεστο είναι ότι έχουμε την μεγαλύτερη ανεργία και στους νέους. Δεν ξέρω στην τελευταία αλλαγή νομίζω Πήρε η Ισπανία την πρωτιά σε αυτό, έγινε μια αλλαγή. Έχουμε δυστυχώς προβλήματα τα οποία αφορούν τη φτώχεια, τη μείωση των εισοδημάτων. Όλα αυτά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Εμείς ως ελληνική πλευρά προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αλλαγές στο σύστημα της οικονομίας των κοινωνικών δομών να τα αλλάξουμε, να τα βελτιώσουμε. Και γι' αυτό θα πω στο τέλος σε σχέση και με την ερώτηση που έκανε ο κύριος Πουπάκης το ζήτημα το οποίο αφορά την αδήλωτη εργασία. Σας είπα ότι η αδήλωτη εργασία και το πιστεύουμε είναι από τις πρώτες προτεραιότητές μας. Είναι το ίδιο σε ειδικό βάρος όσο και οι άλλες προτεραιότητες που θέσαμε, το posting, οι οργανισμοί ε, ε, ε, του εργατικού δυναμικού, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, το ίδιο. Στην Ελλάδα είχαμε πολύ υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας. Το τελευταίο διάστημα αναπτύξαμε με δικές μας δυνάμεις, το επαναλαμβάνω με δικές μας δυνάμεις, καινοτόμα εργαλεία, τα οποία πραγματικά ε, μια πολύ γρήγορη περιγραφή που θα σας κάνω θα σας δείξω ότι είναι καινοτόμα και θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και από άλλες χώρες που δεν λειτουργούν μόνο στη λογική του, ε, της επιβολής των προστήμων, όπως ε, υπόθηκε, αλλά έρχονται και λειτουργούν και θεραπευτικά. Πιάνουν την αδήλωτη εργασία πιο μπροστά. Ε, δημιουργήσαμε το ε, εργαλείο που λέγεται Εργάνη. Ένα εργαλείο το οποίο είναι καινοτόμο, 100% αξιόπιστο, το οποίο απάλαξε από τη γραφειοκρατία όλες τις υπηρεσίες, τις δημόσιες υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας στην Ελλάδα, αλλά και τις, όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ήταν το όφελος των επιχειρήσεων με τη δημιουργία του Εργάνι με το εργάνι πολύ απλά, ανεξάρτητα αν πρόκειται για προσωρινή απασχόληση, έστω και αν είναι δύο φορές την εβδομάδα ή δύο ώρες την ημέρα, η καταγραφή της απασχόλησης γίνεται σε real time υποχρεωτικά από όλες επιχειρήσεις με το πάτημα ενός απλό κουμπιού από την, από την έδρα της επιχείρησης. Καμία σχέση με δήλωση στην, ε, στο, επιθεώρηση εργασίας. Αυτό άλλαξε την εικόνα της Ελλάδος. Σήμερα εγώ ως υπουργό Εργασίας μπορώ και παρακολουθώ όλη την ελληνική οικονομία από το γραφείο μου σε real time ενός δευτερολέπτου. Μπορώ να βλέπω οποιαδήποτε επιχείρηση κάνει πρόσληψη ή απόλυση μερικής, περιοδικής, προσωρινής ή πλήρους εργασίας. Το εργαλείο αυτό είναι στη διάθεση όποιων επιθυμούν να το έχουν. Με αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα είναι απίστευτα θετικά. Όχι μόνο για την καταπολέμηση της αδήλωτης, που πλέον μπορούμε να κάνουμε στοχευμένους ελέγχους, αλλά και γιατί πλέον οι πολιτικές απασχόλησης μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες. Γνωρίζουμε καθαρά την αγορά εργασίας και βλέπουμε τις ανάγκες της. Το επόμενο διάστημα θα αναζητήσω σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις με, μία, με ένα ερωτηματολόγιο να μου καταγράψουν τις ανάγκες τους. Αυτό σημαίνει ότι θα έχω πλέον για πρώτη φορά τόσο αξιόπιστη καταγραφή αναγκών εργασίας. Αυτό το σύστημα εργάνει. Βλέπετε λοιπόν ότι χτυπάει την αδήλωτη. Μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες πολιτικές απασχόλησης και να δούμε και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με αυτό λοιπόν το σύστημα, σε συνδυασμό με το Άρτεμις, το οποίο είπα πριν, με το οποίο πλέον αυστηροποιήσαμε τα πρόστιμα, στην Ελλάδα με λένε υπουργό που έβαλα το υψηλότερο πρόστιμο ιστορικά που μπήκε ποτέ για την αδήλωτη εργασία. Μέχρι πρότινος το πρόστιμο αυτό ήταν 100 ή 200 ευρώ και, τελική, ε, ε, και στο τέλος δεν έμπαινε κιόλα. Ε, έβαλα αυτό το πρόστιμο, το έφτασα σε 10.500 ευρώ και τα πράγματα άλλαξαν. Μέσα από την Εργάνη εκτοξεύτηκε προς τα πάνω το ισοζύγιο προσλήψεων και τα εύσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών τους τρεις τελευταίους μήνες αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια πτώσης. Ε, σαν, για τον κύριο Πουπάκη... Ε, σαν, okay. Και τον κύριο Πουπάκη, ε, κύριε Πουπάκη, να σας πω, πολύ σωστή ερώτησή σας, προτεραιότητά μας είναι το scoreboard. Οι κοινωνικοί δείκτες είναι στις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουμε στην Ελλάδα να κάνουμε κάτι που δυστυχώς δεν το είχαμε μέχρι τώρα, το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, και να κάνουμε και μια αναμόρφωση κοινωνικής πολιτικής μέσα από την πράσινη βίβλο. Αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη. Εννοείται ότι ό,τι είναι στην πρόθεση ε, μιας ενιαίας αντιμετώπισης των ζητημάτων των κοινωνικών δεκτών, θα το προωθήσουμε και θα το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ωραία, λοιπόν. Ε, περνάμε στο δεύτερο γύρο παρεμβάσεων. Η κυρία Μωρά Σαρτιέ και μετά ο κύριο Τούσας. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, που είστε σήμερα εδώ. και που ήρθατε να μας παρουσιάσετε την, το όραμα που έχετε για την Προεδρία σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Εξ ονόματος του ΕΛΚ και του Σάμπα ορι που είναι ο συντονιστής μας και χρειάστηκε να λείψει αλλά και ως μόνιμη συγγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τάμιο θα ήθελα να σας θέσω μια πρώτη ερώτηση. Αναφέρατε το πρόβλημα της ανεργία των νέων που πλήττει ιδιαίτερα τη χώρα σας και ιδιαίτερα ορισμένες περιφέρειες γιατί η ανεργία των νέων φτάνει στο 72% ε, αλλά ε, το πρόβλημα αυτό πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη και γι' αυτό και φτιάξαμε την ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων με ένα άμεσο κονδύλι ε, για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ποια είναι τα μέτρα, τα εφαρμοστικά, ώστε να γνωστοποιηθεί αυτό το front loading, η προκαταβολή δηλαδή ε, χρημάτων και να μπορέσει ε, τα κράτη να το εκμεταλλευτούν και να είναι πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά. Διότι εφόσον καταφέραμε να πετύχουμε το front loading, τώρα πλέον εσείς πρέπει να συνεχίσετε τις ε, κατάλληλες ενέργειες ώστε να υλοποιηθούν όλα αυτά. Δεύτερη μου ερώτηση αφορά την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Μιλήσατε για τον αγώνα σας ε, κατά της ε, μαύρης αγοράς, ε, του κοινωνικού ντάμπινγκ, της παράνομης ή αδήλωτης εργασίας. Για μας εδώ, για όλες τις ομάδες της Επιτροπής μας, η επιτυχία και η οριστικοποίηση αυτής της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους είναι ουσιώδης τη στιγμή που πρόκειται να ξεκινήσουμε την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογέ, διότι η ισχύουσα κατάσταση ε, παίζει υπέρ των ευρωσκεπτικιστών και των λαϊκιστών, πράγμα που όλοι μας θέλουμε να αποφύγουμε φυσικά. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας, ποια είναι η πραγματική σας βούληση για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για αυτή την οδηγία, διότι αυτό που επιθυμούμε εδώ εμείς και ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμή αυτή την, εδώ την Επιτροπή, στόχο είχε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε για την οδηγία στην ολομέλειά μας πριν από τις ευρωεκλογέ. Τέλος, τρίτο μου σημείο αφορά την ε, έκθεση του φίλου και συν, της φίλης και συναδέλφου Ρόδικ Κράτσα. Η, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε σαφή θέση κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του ψηφίσματος στην Ολομέλεια, επιβεβαιώνοντας ε, την ισχυρή του δέσμευση προς μια ισορροπημένη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στις θέσεις κλειδιά των μεγάλων επιχειρήσεων. Η θέση του Ευρωκοινοβουλίου είναι ισορροπημένη και ρεαλιστική και προσφέρει στο Συμβούλιο μια καλή για να μπορέσει να συνεχίσει την εργασία του ε, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία κατά τη διάρκεια της δικής σας ε, ελληνικής προεδρίας. Η κυρία Ρόδη Κράτσα που είναι συνεισηγήτρια της νομοθετικής έκθεσης στο Κοινοβούλιο μου επιβεβαίωσε, με ενημέρωσε μάλλον και εσείς το επιβεβαίωσατε ότι στηρίζετε αυτή την πρόταση. Κατά συνέπεια σας ρωτώ ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Προεδρία ώστε να προωθήσει την ολοκλήρωση ε, της διαπραγμάτευσης για την οδηγία. Σας ευχαριστώ. Έχω πάρα πολλές ελπίδες από την επιτυχία, για την επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας, γιατί αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα της Ευρώπης για, για τους Έλληνες, αλλά και ένα πολύ καλό μήνυμα για το σύνολο των Ευρωπαίων συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα όσα θα κάνετε για να επιτύχετε. Ε, ο κύριος Τούσας, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, έχει προηγηθεί ένα τριήμερο της διακοινοβουλευτικής ε, διάσκεψης μεταξύ των Ευρωβουλευτών και Βουλευτών από τα Εθνικά Κοινοβούλια όπου έχουν κατατεθεί οι πολιτικές προτάσεις και σε ό,τι αφορά το πολιτικό συμπέρασμα που μας αφορά ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θέλουμε να επισημάνουμε ότι στα πλαίσια εφαρμογής της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπη 2020 θα ενταθεί η αντιλαϊκή πολιτική και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας με βασικό στόχο τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης για τη διασφάλιση της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Έχουμε την ετήσια επισκόπηση για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις του 2013 που ανακοίνωσε χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα αξιοποιηθεί και για την προετοιμασία της ετήσιας επισκόπησης για το 2014, για το 2014 στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που αποτυπώνεται σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα των εργαζομένων η ανεργία, η φτώχεια σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την ανεργία καταμετράμε 26.700.000 ανέργους, 120 εκατομμύρια να ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τα όρια της στόχιας. Ε, στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι νέοι άνεργοι. Σε ό,τι αφορά την αδήλωτη εργασία, η ίδια η ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χθεσινή της ανακοίνωση διαπιστώνει ότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα η αδήλωτη εργασία, δηλαδή εκατομμύρια εργαζόμενοι χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, χωρίς ασφάλιση και αυτό αποτυπώνεται στη ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών και ιδιαίτερα με οδυνηρές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων. Δύο είναι τα βασικά εργαλεία που έχουν ως βασικό στόχο τη μείωση της τιμής της εργατικής δυνάμης. Το σύμφωνο για το ευρώ που περιέχει η αμοιβή των εργαζόμενων θα γίνεται σύμφωνα με το κόστος εργασίας αναμονάδα παραγωγής του προϊόντος σε συγκεκριμένο χρόνο και αυτό το κόστος θα αξιολογείται σε σχέση με τους ανταγωνιστές και ανταγωνιστές ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία. Είναι η πρόσφατη απόφαση που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Λευκή Βίβλος για τα δημόσια ασφαλιστικά συστήματα στις 21 Μάη του 2013 που περιλαμβάνονται σαρωτικές αλλαγές. Το κόστος εργασίας όπως γνωρίζετε κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι ίσως έχετε ενημερωθεί και στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια μειώθηκε σύμφωνα με έμπειρους αναλυτές και τελειώνω κυρία 25,6% το εισόδημα των εργαζομένων 28, 38% θέλω την επίγεια σας κύριε Πρόεδρε να υποβάλω μια συγκεκριμένη ερώτηση στον κύριο Υπουργό διάβασα στην εφημερίδα αναυτεμπορική, στην εκδήλωση που έγινε για την ανεργία, ότι μειώσατε ήδη στο τέλος του 2012 τις εργοδοτικές εισφορές κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα και σκοπεύετε με ορίζοντα το 2016 να τις περικόψετε κατά 3,1 μονάδες ώστε να έχετε συσσωρευτική μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θέσει εργασία κατά 30.000. Πρώτο, το πρώτο ερώτημά μου είναι το εξή. Αυτή η περικοπή των, ασφαλι... Ε, εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών θα επιφέρει μία ομοίωση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία που υπολογίζεται στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Από πού αντισταθμιστικά θα την καλύψετε από τα οικογενειακά επιδόματα του ΑΕΔ που παίρνουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ. Και τι αύξηση των... Τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω. Πρόεδρος διακόπτη τον κύριο Τούσα, ο χρόνος σας έληξε. Δεν έχετε πλέον το λόγο. Ο κύριος Δαρδένα. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σα και για την εισήγησή σα. Εγώ θα επανέλθω σε δύο θέματα. Καταρχήν οι δημόσιε υπηρεσίε απασχόληση, για το θέμα για το οποίο είμαι εισηγητής. Ε, και χάρηκα για τα όσα είπατε για την καταπολέμηση τη ανεργία και των, ανεργία των νέων ιδιαίτερα, αλλά και την ανάγκη να ενισχυθεί η συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στι πολιτικέ απασχόληση. Μιλήσατε για τη δημιουργία ε, του δικτύου των υπηρεσιών απασχόληση. και και τις, τα απαραίτητα βήματα για να δημιουργηθεί ένα επίσημο τέτοιο δίκτυο. Εμεί είμαστε πεπισμένοι σε αυτή την Επιτροπή για το ρόλο των δικτύων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόληση όσον αφορά την καταπολέμηση τη ανεργία, αλλά και όσον αφορά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών στο θέμα, αλλά και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, που είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε επιμείνει στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και άρα και στην ανάγκη ανταλλαγή πρακτικών, αλλά και παρακολούθηση του θέματος της υπόθεσης με κατάλληλους δείκτες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό όλα τα κρατημέλη να είναι γύρω από το ίδιο τραπέζι, γύρω από το ίδιο δίκτυο και μόνο αυτή η προϋπόθεση θα δώσει μια πραγματική προστιθέμενη αξία στα επίσημα αυτά δίκτυα των δημοσίων υπηρεσιών απασχόληση. και μιλούσατε για προαιρετικό χαρακτήρα. Χθε προσπαθήσαμε να επιδείξουμε δημιουργικότητα με τους εκπροσώπους σας για να βρούμε κάποια λύση. Και από ό,τι κατάλαβα, ήμασταν σύμφωνοι ως προς αυτό, αλλά ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να έχω την συγκεκριμένη τη δική σας γνώμη. Δεύτερο σημείο που είναι ανεξάρτητο από το το είναι το να επανέλθουμε στην ανάγκη της καταπολέμησης αδήλωτης εργασίας, γενικότερα κατά της κοινωνικής απάτης και κάτι που δεν είναι τελείως ανεξάρτητο και της απάτης, Αν και ξέρουμε πως η Ένωση έχει περιορισμένες αρμοδιότητες στο θέμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή πλατφόρμα για ανταλλαγή πρακτικών, πληροφοριών και νομοθεσιών. Αλλά δεν πρέπει να χάσουμε το στόχο. Θα πρέπει η καταπολέμηση της κοινωνικής απάτης να μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε τις διευθυντικές απάτες των επιχειρήσεων που συχνά οδηγούν σε, σε θυματοποίηση των εργαζόμενων με, εκμετάλλευση διαφόρων ε, νομοθεσιών και παραθύρων αυτών. Σας ευχαριστώ. Ε, Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσατε να απαντήσετε σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις και μετά σας μένω άλλες δύο συν τη δικιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την κυρία Μωρέν Σαρτιέ, ε, ακούσατε και πριν στην ε, τοποθέτησή μου για τις προτεραιότητες ότι το ζήτημα το οποίο αφορά το posting είναι βασική προτεραιότητα. Έχει εκφραστεί σε 9 Δεκεμβρίου η πολιτική βούληση στο ΕΠΣΚΟ και αυτό θέλουμε να το ολοκληρώσουμε μέσα στην ελληνική προεδρία. Με ρωτήσετε για το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα 8 τριλόγων που έχουν ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνονται στις 18 Φεβρουαρίου. Όπως είπα τόσο η απόφαση του Συμβουλίου στις 9 Δεκεμβρίου όσο και του Κοινοβουλίου δείχνει ότι υπάρχει εκφρασμένη πολιτική βούληση. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχάσουμε και δεν πρέπει να χάσουμε. Στόχος μας είναι να αναλάβουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε μέχρι τις 18 Δευτέρου να πετύχουμε τη συμφωνία που είναι και το ετούμενο των λαών της Ευρώπης. Το είπα και πριν και το επαναλαμβάνω. Γνωρίζω ότι το εγχείρημα είναι δύσκολο διότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Όμως αυτή είναι η δύναμη της Ευρώπης, η σύνθεση, η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και προτάσεων. Γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί. Για το ζήτημα της πρωτοβουλίας ε, για τους νέους, για την ανεργία των νέων. Ε, σαφέστατα γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή η το όνομα κρίση, η κρίση στην Ευρώπη έχει όνομα και επίθετο. Λέγεται ανεργία και ανεργία των νέων και εκεί πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Και γι' αυτό και αυτό, αυτή την περίοδο, είναι μέσα στις βασικές μας προτεραιότητες. Η πρωτοβουλία για την, ενασχόληση, για την απασχόληση λοιπόν των νέων είναι κεντρική προτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία. Θα αξιολογήσουμε τα εθνικά προγράμματα τα οποία έχουν υποβληθεί μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτου και οι πρώτοι απολογισμοί θα παρουσιαστούν στο έψικο του Ιουνίου. Στις 8 Απριλίου θα λάβει η χώρα ένα σημαντικό συνέδριο υπό την αιγίδα της Προεδρίας και της Επιτροπής, στο οποίο θα συμμετέχει και ο ίδιος Πρωθυπουργός χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς, γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα, δείχνοντας το ενδιαφέρον και το ειδικό βάρος που δίνουμε στο θέμα της ανεργίας των νέων. Για τον κύριο Νταρνέν, για το δίκτυο δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Ε, είμαστε πράγματι κοντά σε συμφωνία, αυτή είναι η εκτίμησή μας θέση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου δεν είναι πλέον μακριά οι θέσει Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Τα κράτη-μέλη πιστεύουν στη συμβολή και την προστιθέμενη αξία αυτού του δικτύου. Για το λόγο αυτό άλλωστε εξέδωσαν και δήλωση που εκφράζουν ακριβώς τη βούλησή τους για την αξιοποίηση αυτού του δικτύου. Ε, με λίγα λόγια πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ε, λύση, θα υπάρξει συμβιβασμό. Και αυτό είναι που μας δίνει τη χαρά και την ελπίδα ε, ότι θα γίνει πολύ σύντομα. Ε, για το θέμα της, ε, του κυρίου ε, Τούσα. Πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Το ξέρετε, στο πλαίσιο μεγάλων και σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Και η προσπάθεια αυτή στην καταπολέμηση και της ανεργίας, η οποία δεν λύνεται η ανεργία και αυτό το ξέρουμε ούτε με νομοθετήματα, ούτε με νόμους, ούτε με ευχές. Η ανεργία αντιμετωπίζεται με ανάπτυξη. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλάζουμε και στο labor market παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. Μία από αυτές ήταν ότι δυστυχώς είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα μη μισθολογικά κόστη στην Ευρώπη. Γι' αυτό στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και αυτό που έκανα και εγώ ως υπουργό ήταν καταρχήν να μειώσουμε κατά μία ακόμα μία μονάδα που είναι σημαντική μείωση το μη μισθολογικό κόστος. Και στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2016 να μειώσουμε κατά 3,9 μονάδες συνολικά 5. Αυτή η μείωση είναι πάρα πολύ σημαντική για την προσέλκυση επενδύσεων, γιατί μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων θα έρθει ανάπτυξη και μέσα από την ανάπτυξη θα χτυπήσουμε και το νοσηρό φαινόμενο της ανεργίας. Αυτή είναι η οπτική της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι η λογική οπτική. Γιατί υπάρχει και η άλλη οπτική. Η άλλη οπτική που παντού θέλει να κάνει να εργάζονται όλοι, που το θέλουμε όλοι αυτό, αλλά με ποιου πόρου, μαγικούς. Υπάρχει κάποιο που γνωρίζει ένα κουμπί που αν το πατήσουμε μπορεί αυτόματα να απασχοληθεί το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών ανέργων που έχουν ανάγκη των νέων. Όχι. Αυτό γίνεται με προσπάθειες, με ανταγωνισμό, με ανάπτυξη. Σε αυτή την κατεύθυνση η ελληνική κυβέρνηση είναι προσιλωμένη και κάνει συγκεκριμένα βήματα τα οποία δείχνουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, But then it means he has nothing to answer to you. Για να μην σας απαντάει, μάλλον δεν έχετε να σα πει. Σάρι Εσάια και μετά η κυρία Μπεναμπάρ Ατού. Ευχαριστώ. θα έχετε και άλλη ευκαιρία για συνέχεια της συζήτησης. Ούτως ή άλλως ε, αγορεύσετε αρκετή ώρα. Οπότε από σεβασμό προς τα άλλα μέλη ας μην ε, παρατείνουμε αυτή τη διμερή συνομιλία με τον Υπουργό. Κυρία Σάια, συμφωνώ μαζί σας κυρία Πρόεδρε ότι θέμα της συζήτησης είναι η προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, όχι η εσωτερική ελληνική συζήτηση. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας. Στην Επιτροπή μας εξετάσαμε πολλές οδηγίες και προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που δημιουργεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασυνοριακά αλλά και από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μωράν Σαρτιέ σας μίλησε για το χρονοδιάγραμμα της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων και ευχαριστώ για την απάντηση που δώσατε. Θα ήθελα τώρα να μα παρουσιάσετε το χρονοδιάγραμμα για την οδηγία ICT, γιατί αυτή έχει κολλήσει κάπου στον τριμερή διάλογο. Έχουμε και την οδηγία για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως φοιτητές ή ερευνητές και τους ασκούμενους ε, είτε έχουν αποδοχές είτε όχι. Υπάρχει δυνατότητα και αυτές τις σημαντικές οδηγίες να τις διεκπαιρεώσουμε στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Γιατί δεν υπάρχει οδηγία που να είναι παρόμοια με αυτές τις δύο. Είχαμε μία άλλη οδηγία που ολοκληρώθηκε πριν το Δεκέμβριο και θα περάσει την Ολομέλεια το Φεβρουάριο για τους εργαζόμενους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, παρατηρείται, θα έλεγα, μία ξενοφοβική, ένα ξενοφοβικό, για να μην πω ρατσιστικό ύφος στη συζήτηση. Έχετε κάποιες ε, ιδέες, κάποιο σχέδιο για το πώς θα γίνει η συζήτηση αυτή στα πλαίσια και της προεκλογικής εκστρατείας, ώστε να κατευναστεί κάπως αυτό το έντονο ξενοφοβικό ύφος και να προσαρμόζεται σε πραγματικά στοιχεία και περιστατικά. Γιατί γνωρίζουμε από μελέτες ότι λιγότερο από 3% του εργατικού δυναμικού εργάζονται σε άλλες χώρες μέλη. Οπότε δεν υπάρχει λόγος για τέτοιες δηλώσεις ξενοφοβικές. Η κυρία Μαλίκα Μπεναμπάρ Ατού. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, στην ε, αρχή της ομιλίας σας μιλήσατε για το κίνδυνο της ανόδου του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού. Όντως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και πολύ συχνά στις συναντήσεις ε, με τους συμπολίτες μας ακούμε την περίπτωση της Ελλάδας, γιατί υπάρχει κρίση, αλλά και ε, έχουμε και την Τρόικα που απέτησε μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν σε μεγαλύτερη φτώχυνση του πληθυσμού. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του τι απέφχονται για την Ευρώπη οι Ευρωπαίοι πολίτες. Επίσης μιλήσατε για τα νέα εργαλεία που έχετε προκειμένου να αποκομίσουμε καλύτερες γνώσεις για την κατάσταση αγοράς εργασίας. Η επενδυτική πολιτική αφορά περισσότερο μεσοπρόθεσμες πολιτικές, ενώ έχουμε άμεσες απαιτήσει και ανάγκες. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν ήδη από τώρα, και θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε, να ε, προσαρμόσουμε την ευρωπαϊκή συζήτηση και στο παγκόσμιο προσκήνιο, γιατί στην, στον έχουμε μια επιτροπή, την Επιτροπή Μπασιλέ, που ζήτησε την συμπερίληψη του κοινωνικού πυλώνα και στις παγκόσμιες συζητήσεις. Γιατί στην αρχή η συζήτηση αυτή αναφερόταν μόνο στις φτωχότερες χώρες, στις χώρες του Νότου. Αλλά διαπιστώνω ότι σήμερα ήδη στην Ευρώπη έχουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα πυλώνα κοινωνικής προστασίας, ώστε να δώσουμε σε όλους τους συμπολίτε μας την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην υγεία, η ατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε μια αξιοπρεπή σύνταξη για να αποκτήσει τα βιοποριστικά μέσα και ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Συμφωνείτε με την ιδέα αυτή να δώσουμε ένα τέτοιο πυλώνα κοινωνικό και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι συναφής με την ερώτηση της κυρίας Μπεναμπάρα του και με, την κοινοβουλευτική εβδομάδα που έχουμε και τις συνομιλίες με τις εθνικές βουλές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση για την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Από πολλά συμπεράσματα του Συμβουλίου δυστυχώς φαίνεται ότι δεν είναι προτεραιότητα το θέμα αυτό για το Συμβούλιο. Προτεραιότητα για το Συμβούλιο είναι αυτά τα περίφημα συμβόλαια. Συμβόλαια όμως που θυμίζουν κάποια ήπια τρόικα. Δεν είναι τα συμβόλαια αυτά, τις συμβάσεις αυτές, προσπάθεια μέρημνας για σημαντικές πτυχές της αλληλεπίδρασης που υπάρχει γιατί υπάρχει επίδραση που δείχνει ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρο την κοινωνική διάσταση και τις κοινωνικές πτυχές. Και δυστυχώς ε, υπάρχουν ανισορροπίες στα δημόσια οικονομικά, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέπουμε το κοινωνικό θέμα. Πώς βλέπετε λοιπόν ε, τη μερίσια διάταξη του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόληση ΕΠΣΚΟ, γιατί φαίνεται να απουσιάζει από τα συμπεράσματα το κάτι τέτοιο. Βέβαια, Έχουμε επιτάπητο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως είναι αποσπασματική και αφορά μόνο τους δείκτες. Για τους δείκτες κατάλαβα, αντιλήθηκα ότι θα ασχοληθείτε και, θα, με τους δείκτες θα ασχοληθείτε κι εσείς. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και πολλά εθνικά κοινοβούλια, επιμένουμε να προσθεθούν και άλλοι δείκτες. Πέραν του δημογραφικού δείκτη, το θέμα της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, άστεγη, φτώχεια των παιδιών. Και επιμένουμε να συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι σε αυτόν τον κοινωνικό διάλογο. Το θέμα όμως των δικτών δεν εξαντλεί τη συζήτηση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τους αξιοποιήσουμε, πώς θα τους χρησιμεύσουμε. Ούτε παραλαμβάνω εξαντλείται το κοινωνικό ζήτημα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ με τους δείκτες. Στην Επιτροπή μας οργανώσαμε τον Ιούλιο μια πολύ σημαντική δημόσια ακρόαση με θέμα την θέσπιση μιας ελάχ... ενός ελάχιστου επιδόματος ανεργίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι αυτή η συμβολή, στη δημιουργία ενός ε, αυτόματου σταθεροποιητή, τουλάχιστον στην Ευρωζώνη, είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν μπορώ να σας αναπτύξω όλους εδώ. Δεν έχω το χρόνο. Θα ήθελα πάντως ε, αυτό να επαληθεύσω με την Ελληνική Προεδρία, ότι μένουν ανοιχτέ αυτές όλες οι προοπτικές ε, για συζήτηση. Γιατί αν συνεχίσετε να συζητάτε το θέμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώνει τη θητεία του και δεν θα είμαστε εκεί για να σας δίνουμε κάποιες ενδείξεις. Τώρα, πάνω κάτω στο ίδιο θέμα, έχω και μια δεύτερη ερώτηση, αλλά υπό διαφορετικό πρίσμα. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και όχι μόνο, και στα δικά μας ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε στο blueprint, είτε στην ανακοίνωση του Οκτωβρίου, έχουμε το θέμα του κοινωνικού διαλόγου και τις θέσεις που θα πρέπει να έχει ο κοινωνικός διάλογος. Εγώ λέω ότι η συζήτηση αυτή είναι πολύ... είναι για τα μάτια ουσιαστικά. Απλώς λέμε το όνομα και θεωρούμε ότι έτσι εξαντλήσαμε τη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση ουσιαστικά συμβολική. Τώρα, δεν ξέρω πότε θα γίνει τριμερής αυτή η κοινωνική σύνοδος κορυφής. Όλα αυτά είναι πολύ πιο τυπικά και επίσημα. Και οι χώρες που έχουν επιτυχία στη μεταρρυθμίση είναι αυτές που έχουν κοινωνικό διάλογο και λειτουργούν εύρυθμα. Εμείς ε, λυπούμαστε που στην Ελλάδα η επέμβαση της Τρόικα, που μάλιστα καταγγέλθηκε και από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και από το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, ουσιαστικά αρνείται τα ίδια τα θεμέλια της συλλογικής διαπραγμάτευσης αλλά εμείς διαρωτόμαστε πώς μπορούμε να ανανεώσουμε, να αναπτύξουμε, να αναζωογονήσουμε αυτό το κοινωνικό διάλογο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί οι ανισορροπίες που διαπιστώνουμε σε κοινωνικό επίπεδο θα πρέπει να συζητηθούν με συμμετοχή όμως των κοινωνικών εταίρων. Για να είναι αμφίδρομη η πορεία και για να συμβάλλουν οι κοινωνικοί εταίροι στη συζήτηση αλλά και για να μπορέσουν να κάνουν κτήμα τους στα συμπεράσματά, στα συμπεράσματά σας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι λοιπόν που συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μέχρι στιγμής όλα παραμένουν σε τυπικό και συμβολικό επίπεδο και όχι στην ουσία. Αυτές ήταν οι μου κύριε Υπουργέ και σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε στις τρεις τελευταίες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να ξεκινήσω από τις παρατηρήσεις παύλα ερωτήσεις της Προέδρου της κυρίας Μπέρες και να πω ότι μέσα μας βαθιά γνωρίζουμε την αναγκαιότητα λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης που υπήρξε στην Ευρώπη ότι έπρεπε να υπάρξει δημοσιονομικός εξορθολογισμός, δημοσιονομική εξυγίανση αλλά και δημοσιονομική προσαρμογή σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις όπου ήταν αναγκαίες, σε όποιες χώρες. Όμως, το έχω πει με την ευκαιρία συζητήσεων και στο ΕΠΣΚΟ, αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή ποτέ δεν ήταν και δεν πρέπει να είναι ο αυτοσκοπός. Αυτοσκοπός για την Ευρώπη και τις χώρες είναι αυτό που λέγεται κοινωνική συνοχή και κοινωνική ευημερία. Το μέσο και το εργαλείο είναι η δημοσιονομική προσαρμογή για να φτάσουμε σε αυτό που είναι η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ευημερία. Αυτό είναι ο στόχος. Η κοινωνική Ευρώπη, η ευτυχία στους πολίτες, η αύξηση του βιωτικού επίπεδου. Η δημοσιονομική προσαρμογή, κυρία Πρόεδρε, είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε εκεί. Αυτά τα δύο λοιπόν συνδέονται και βρίσκονται σε μια ισορροπία. Μια ισορροπία εύθραστη, την οποία πρέπει να τηρήσουμε. Και αυτός πρέπει να είναι ο κοινός μας στόχος. Το ζήτημα το οποίο αφορά την κοινωνική διάσταση όσο αφορά τους δείκτες. Ε, εγώ γνωρίζω ότι πολλά πράγματα, και έτσι γίνεται, δεν γίνονται με άλματα, αν και θα έπρεπε ίσως. Γίνονται όμως με σταθερά βήματα. Το ότι προχωράμε τώρα σε αυτό το εξάμεινο, στην κατάκτηση κάποιων πρώτων κοινωνικών δικτών που λέγεται scoreboard, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Εννοείται ότι αυτό δεν μπορεί να το πει κάποιος τέλειο. Και εννοείται ότι σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτά που χθε είπατε και συμφωνώ απόλυτα και άλλους κοινωνικούς δείκτες και αυτόν που είπα από πλευράς της, της Ελλάδος για το δείκτη της δημογραφικής καταγραφής για μια Ευρώπη που γερνάει, το δείκτη για τη φτώχεια των παιδιών, το δείκτη της υγείας. Κανείς δεν έχει αντίρρηση με αυτό. Αλλά το θετικό είναι ότι πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα. Και το πρώτο βήμα γίνεται. Γίνεται η πρώτη καταγραφή πλέον κοινωνικών δικτών. Και είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό πρέπει να το εχαιρετήσουμε και να το στηρίξουμε. Και έχουμε όλο το χρόνο, εμείς ή οι επόμενοι από εμά, να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Και έτσι γίνεται στην Ευρώπη. Από γενιά σε γενιά, από συμβούλιο σε συμβούλιο, από κοινοβούλιο σε κοινοβούλιο έρχονται και προστίθενται συνεχώς νέες προτάσεις, ιδέες, αξίες που δυναμώνουν το ευρωπαϊκό όραμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι αισιόδοξο ότι αυτό θα προχωρήσει. Για τον κοινωνικό διάλογο. Πράγματι, ο κοινωνικός διάλογος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν είναι το ίδιο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ως θεσμός κατοχυρωμένος. Και στην Ελλάδα έχουμε προβλήματα στον κοινωνικό διάλογο. Και δεν ήταν αποτέλεσμα της Τρόικα. Ήταν ένα έλλειμμα οριμότητας που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία όσο αφορά το διάλογο πολύ πριν την Τρόικα. Και αυτό προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Και ξεπερνάμε την Τρόικα γιατί το θέλουμε να το κατακτήσουμε και αυτό πρέπει να γίνει κτήμα για όλη την Ευρώπη. Πράγματι, ο διάλογος έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αν και είναι στα πρώτα του στάδια, γιατί είναι στα πρώτα του στάδια, έχει θέσει ήδη σοβαρά ερωτήματα όπως είναι για την εισαγωγή μηχανισμού αυτόματος σταθεροποιητών. Ε, αυτό το διάλογο η Ελληνική Προεδρία έχει σκοπό να τον εξετάσει στο πλαίσιο του άτυπου ΕΠΣΚΟ στην Αθήνα 29 και 30 Απριλίου. Αυτό είναι μια ημερομηνία στο χρονοδιάγραμμα για τον κοινωνικό διάλογο. Θα σας πω ότι η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, γιατί έχει αξία να το πούμε αυτό, πριν ένα μήνα, στο, στο επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου, συμφώνησε μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους συμφωνία κλαδική μέσα στη, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και του μνημονίου που έδινε αύξηση μισθού, που σημαίνει ότι οι ελπίδες υπάρχουν. Ε, το σχέση με που Ε, για το θέμα, ε, για το άλλο θέμα είναι ότι θα εργαστούμε για να ενσωματώσουμε τα θέματα των ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο του διαλόγου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την αναπτυξιακή διάσταση της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020. Και νομίζω ότι εκεί είμαστε. Ε, για αυτό που είπε η κυρία Εσάγη για το πρώτο, είναι ότι ε, τα πρώτα που ακούστηκαν είναι, δεν είναι απασχολούν και δεν είναι αρμοδιότητά μας. Όμως η Ελληνική Προεδρία στην ε, αρμόδια σύνθεση του Συμβουλίου καταβάλει κάθε προσπάθεια και ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρξει πρόοδος. Δεν υπάρχει. Ε? ε αυτό. Euh, Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρίγνερ έφτασε καθυστερημένη. Είχα κλείσει τον κατάλογο μιλητών. Δεν υπάρχει λόγο να σα δώσω το λόγο εγώ. Αλλά επειδή έχουμε λίγο χρόνο, σα προτείνω παρόλα αυτά να του δώσουμε το λόγο. Να της δώσουμε το λόγο. Και κατάλαβα και ότι ο Αλεχάνδρο Σέρκα θέλει να πάρει και εκ νέου το λόγο. Υπάρχει κάποιο άλλο, Όχι. Ωραία λοιπόν η Εύελιν Ρέγνερ, μετά ο Αλεχάνδρο Σέρκα και μετά θα ολοκληρώσουμε, κύριε Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η ερώτηση που επιθυμώ να θέσω, αρχικά την έθεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνη και γι' αυτό δεν ήμουν και έγκαιρα εδώ. Με ενδιαφέρει το θέμα της εξισορροπημένης σχέση ανδρών και γυναικών στις εποπτικά συμβούλια. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή η, έχει συνταχθεί έκθεση από την Νομική Επιτροπή αλλά και από την Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών και θα εγκριθεί από τους Υπουργούς Κοινωνικών Υποθέσεων. Εγώ δεν είχα ωστόσο την ευκαιρία μέχρι τώρα να λάβω απάντηση στην ερώτησή μου, διότι προφανώς οι αρμοδιότητες των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι διαφορετικές από την κατανομή των αρμοδιοτήτων στο Συμβούλιο. Γι' αυτό η ερώτησή μου είναι ποια στάση θα τηρήσει η ελληνική προεδρία για το θέμα αυτό. Θα, θα προσπαθήσει να επιτελέσει κάποιε προόδου. Συγγνώμη που εκνευρίζομαι, αλλά Εάν φτάσατε αργά, ένδειξε δεν ενημερώνεστε γιατί είπε ο υπουργό. Στην εισαγωγική του ομιλία ανέφερε και αυτά τα θέματα. Λυπάμαι, ε, εκνευρίζομαι, αλλά θα πρέπει να ενημερωνόμαστε. Από τη στιγμή που δεν ερχόμαστε εγκαίρως, τουλάχιστον να, να ενημερωνόμαστε για το τι υπόθηκε πριν από εμά, για να μην ε, υποβάλλουμε τέτοιε ερωτήσει. Εγώ ήμουν, δεν είμαι εδώ, αλλά έκανα τέτοιε ερωτήσει. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν κάποιε φήμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυκλοφορούν κάποιε φήμε ότι ετοιμάζεται αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ώστε να αποκλειστεί μια δυσάρεστη εικόνα για τους υπουργούς, ε, για, το... για να μην φανεί ότι η... ο στόχος εξάλληψης φτώχειας αντί να υλοποιείται στην Ευρώπη φαίνεται ότι η κατάσταση της φτώχειας επιδεινώνεται. Μπορείτε να σταθείτε στο πλευρό μας ώστε αυτές οι φήμες να μην υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. J'ajoute à l'intervention να προσθέσω κι εγώ σε αυτά που είπε ο κύριος Σέρκας, ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε βέβαια κάποια συλλογική απόφαση, αλλά το να διορθώνει η απερχόμενη ε, Επιτροπή αυτή τη στρατηγική και να μην ε, δίνεται ευκαιρία στο νέο Κοινοβούλιο και στη νέα Επιτροπή με την νέα εντολή της να επεξεργαστούν τα θέματα αυτά είναι θέμα πολύ σημαντικό και είναι και μίζουν ε, ένα πολιτικό μήνυμα που θα μπορούσε να δώσει εδώ η ελληνική προεδρία. Και από άποψη Δημοκρατικής Λειτουργίας Ένωσης ήταν κάτι πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στην κυρία Ρένκερ, παρότι, όπως είπατε, δεν άκουσε την ε, εισήγησή μου. Διαβάζω από το κείμενο της εισήγησής μου, κυρία Ρέγκερ, ότι εντός των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας συμπεριλαμβάνεται το ζήτημα των ίσων ευκαιριών και της μάχης κατά των διακρίσεων. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, η ελληνική προεδρία θα συνεχίσει την εξέταση της πρότασης για μια οδηγία για την ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την πίστη, την αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό Επιπλέον θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης της πρότασης για μια οδηγία για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών που είναι εγγεγραμμένες στο χρηματιστήριο. Άλλωστε το θέμα από ελληνικής πλευράς είναι πολύ γνωστό γιατί το έχει αναδείξει πολύ εύσοχα και έντονα η κυρία Κράτσα με την οποία έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Όσο για το θέμα ε, που έθεσε ο αγαπητός ο κύριος Σέρκας. Η Επιτροπή αναμένεται να δημοσιοποιήσει έκθεση απολογισμού για την Ευρώπη 2020. Αυτό το σενάριο δεν υφίσταται για την εξαίρεση του στόχου για τη φτώχεια. Αυτό είναι που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Monsieur le Ministre. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Στο όνομα ε, του συνόλου των μελών ε, της Επιτροπής ε, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και όσων έμειναν μέχρι το τέλος, σας ευχόμαστε καλή δύναμη για την Προεδρία σας και για όλες αυτές τις νομοθετικές βάσεις που πρέπει να ολοκληρώσετε. Στην ίδια βάρκα είμαστε όλοι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να την κυβερνήσουμε μαζί για να φτάσουμε σε αίσιο πέρα. σα ευχαριστώ λοιπόν. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίε μας. Θα τα ξαναπούμε στις 3 Φεβρουαρίου στην έκτατη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο στις 7 η ώρα το απόγευμα.